Chers collègues, je vous propose de prendre place pour que nous puissions. Είμαστε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Ο κύριος Τόμας Μάν. Äh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χθε υπήρξε μια μεγάλη διαδήλωση στις ε, Βρυξέλλες από τους ε, ε, συναδέλφους που απασχολούνται στις κατασκευές στην Γερμανία. Ξέρω ότι βέβαια είναι θέμα δικαίου ανταγωνισμού, ε, το ότι θέλουν να κλείσουν κάποιες επιχειρήσεις στην, ε, τέτοιες στην ε, Γερμανία, αλλά εμείς ως Επιτροπή για την Απασχόληση ποιες δυνατότητες έχουμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Σήμερα θα κλείσουν κάποιες τέτοιες επιχειρήσεις στην Γερμανία διότι έχουν καταργηθεί κάποια επιδόματα. Αυτό μπορεί να πλήξει και άλλου ε, συναδέλφου σε άλλα κρατημέλη. Εμεί ποιε δυνατότητε έχουμε ω Επιτροπή Απασχόληση να ασχοληθούμε με το θέμα. Κυρία Πρόεδρε, και εγώ γνωρίζω εκ του αυτή την κατάσταση η οποία πλήττει συγκεκριμένες ε, ισπανικές ε, περιοχές και έχει και μία πάρα πολύ βαριά κοινωνική επίπτωση που θα μπορούσε να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο λαό. Ο πληθυσμός είναι απελπισμένος και είναι απελπισμένος διότι διαπιστώνει ότι στην Ευρώπη δεν είναι πρώτο μέλημα η απασχόληση, ίσα ίσα βρίσκεται στο τέλος. Ανησυχεί για την οικονομία, αλλά ο κόσμος είναι απελπισμένος. Και καλό θα ήταν να ακούσουμε τουλάχιστον αυτούς τους ανθρώπους. Θα έπρεπε να τους δώσουμε τη δυνατότητα, δεν ξέρω, να κάνουμε μια ακρόαση εδώ στην Επιτροπή μας, ώστε να εισακουστούν. Διότι αυτή τη στιγμή νιώθουν ότι τους αγνοούν και προέχουν τα συμφέροντα ε, χωρών ε, που έχουν ε, και γίνονται εισαγωγές από χώρες που έχει μικρό εργατικό κόστος, μικρούς μισθούς και ποια είναι η εναλλακτική λύση. Τους αφήνουμε χωρίς ελπίδες, χωρίς μέλλον και χωρίς ε, θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμας Μαν αναφέρθηκε στη διαδήλωση που έγινε χθες. Πολύ γνωρίζετε, το είπε και η κυρία Φέγγερα εχθές, ε, η διαδήλωση που έγινε εχθές είχε πολύ μεγαλύτερη θεματολογία και αφορούσε το σύνολο των θεμάτων που ασχολούν την Επιτροπή Απασχόλησης, ε, ε τα μέτρα λιτότητας τα οποία εφαρμόζονται στη μία στην άλλη χώρα και προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται και με ε, τα χρέη και ούτω καθεξής. Δεν θα ήθελα να ξεκινήσω εδώ μια συζήτηση επικυρεότητας επί του θέματος. Προτείνω στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να είμαστε και εμείς συντονισμένοι με αυτές τις ανησυχίες διότι φυσικά όλα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο της δικής μας εντολής και υπάρχουν μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν να ε, συντονιστούμε και να τα συμπεριλάβουμε στην μερίσια μας διάταξη. Να σας υπενθυμίσω ότι ο Επίτροπος Άντορ θα είναι εδώ σε λίγο για να συζητήσει για το πρόγραμμα εργασίας του, του 2011, αλλά γνωρίζουμε ότι στη συνεδρίαση που έγινε χθε, ε, μια συνεδρίαση που κράτησε πάρα πολύ ώρα, ε, συζητήθηκαν επί τρει ώρες τα θέματα της απασχόλησης. Η ε, συνεδρίαση για τους Ρωμά διέρχεσε δύο ώρες και το θέμα που είπε ο κύριο Μαν ήταν θέμα της συνεδρίασης. Θα το συζητήσουμε και με τον Επίτροπο εντό ολίγου και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό και στις συνεδρίες των συντονιστών. Να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη, να δώσω το λόγο στην κυρία Άρκιν για να μας παρουσιάσει τη γνωμοδότησή της για το ΑΕΠ και πέρα από αυτό τη μέτρηση της πρόοδου σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι είναι το ΑΕΠ. Με μια πρόταση είναι μια περιγραφή του συνόλου της εθνικής παραγωγής, διότι αποτελεί ένα σύνολο των ε, αξιών, των ε, ποσών που έχουμε παράξει. Ε, δεν θα σταθώ περαιτέρω στο ΑΕΠ, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και αν ε, πάμε πίσω στη δεκαετία του 70 που δεν υπήρχαν στοιχεία για να μετρήσουμε τι ακριβώς συνέβαινε με την οικονομία, ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και είναι ένα συνολικό εργαλείο μέτρησης της οικονομικής δραστηριότητας. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος άλλαξε έκτοτε και φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο η κοινωνία αλλά ο ίδιος ο κόσμος άλλαξε και αυτά που αξιολογούμε και τα πράγματα στα οποία προσδίδουμε αξία άλλαξαν. Και επιπλέον το ΑΕΠ πολλές φορές δίνει θετικά στοιχεία ή ε, ε, μετράει θετικά για πράγματα τα οποία ε, ε, για μας είναι καταστροφή. Για παράδειγμα, αν υπάρξει μια καταστροφή, το ΑΕΠ αυξάνεται γιατί λόγω της καταστροφής έχουμε νέα παραγωγή και νέες κατασκευές ή αν κόψουμε πολύ ξυλία από τα δάση, ναι μεν αυξάνεται το ΑΕΠ γιατί έχουμε περισσότερη ξυλία, αλλά ο πλανήτης καταστρέφεται. Σίγουρα λοιπόν το ΑΕΠ δεν, καταστρέφει τον, δεν περιγράφει τον κόσμο όπως τον γνωρίζουμε. Ε, αλλά με κάποιο τρόπο ανταποκρίνεται στις αλλαγές. Μια δεύτερη παρατηρήση που θα ήθελα να κάνω και έχει σχέση με αυτό που συζητούσαμε πριν από λίγο, είναι ότι οι καλές ε, αποφάσεις πολιτικής ε, εξαρτώνται από τις ολοκληρωμένες λύσεις. Αν δεν έχουμε καλές πληροφορίες, δεν μπορούμε να ετοιμάσουμε καλές πολιτικές προκειμένου να ανταποκριθούμε στην τρέχουσα κρίση, επί παραδείγματι. Όταν λοιπόν αναφέρομαι στο ΑΕΠ, δεν αναφέρομαι μόνον στην ακρίβεια των πληροφοριών ή στην ποιότητα των πληροφοριών, διότι είναι ακριβή συνήθω οι πληροφορίε και μια κάποια προϊόντα την έχουν. Μπορεί όμω τα ακριβή στοιχεία να μην περιγράφουν την κατάσταση. Περιγράφουν την κατάσταση μόνο από οικονομική πλευρά και μπορεί να είναι ακριβή μεν από κοινωνική πλευρά, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη του θέματα όπω η βιωσιμότητα, η ευημερία κ.ο.κ. Και επειδή ακριβώ ε, το ΑΕΠ είναι ένα οικονομικό στοιχείο, κατά πάσα πιθανότητα δεν περιλαμβάνονται όλες αυτές οι πολιτικές που είναι καλές για την ευημερία μας και ε, οι πολιτικές οι οποίες ε, ε, οδηγούν στην αύξηση του ΑΕΠ. Υπάρχει και ένα χάσμα μεταξύ του ΑΕΠ και του τρόπου που ο καθένας αντιλαμβάνεται τις συνθήκες τις οποίες βιώνει. να σας επαναλάβω ότι γίνεται σε μια καταστροφή. Το ΑΕΠ αυξάνεται, αλλά η ζωή για τον πληθυσμό και για την κοινωνία ε, είναι πληγμένη. Υπάρχει και διαφορά μεταξύ του του εθνικού εισοδήματο και του καθάριστου εγχώριου εισοδήματο. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε εδώ, αλλά για τη χώρα μου έχει μεγάλη σημασία. Ορισμένε φορέ όμω δίνω μια λανθισμένη εικόνα του τι συμβαίνει. Ο λαός βλέπει τις εικόνες αυτές και τα στοιχεία αυτά και θεωρεί ότι δεν δείχνουν μια καλή εικόνα τη ζωή μου και θεωρούν ότι το ΑΕΠ δεν του αντιπροσωπεύει γιατί αναφέρεται μόνο σε οικονομικά στοιχεία, ε, στη, αναφέρεται μόνο στην αγορά και στις οικονομικέ συναλλαγέ. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε μια δέσμευση προς τους πολίτες ώστε να έχουμε δείκτες ε, που περιλαμβάνουν πιο πολύ τα στοιχεία, να υπάρξει περισσότερη δημόσια ε, συζήτηση και να γίνει καλύτερη χάραξη πολιτικής. Και επίση δεν χρειάζεται να μετράμε μόνο την ποσότητα αλλά και την ποιότητα. Όχι μόνο τι κοστίζει αλλά και τι είναι καλό. Όχι μόνο το κόστος αλλά και την αξία του. Ε, πρέπει να δούμε και τις απώλειες και τα κέρδη. Και έτσι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε και ε, βιωσιμότητα. Την ποιότητα ζωή την ανέφερα, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Πρέπει να δούμε και την πρόοδο, η οποία είναι πολυδιάστατη και δυναμική. Υπάρχουν και δύο-τρία πράγματα που είναι πολύ σημαντικά και θα τελειώσω με αυτά. Θέματα κατανομή. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Διότι η εφημερία μια κοινωνία εξαρτάται και από τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα στοιχεία τα οποία αποτελούν τη ζωή ενό ανθρώπου κατανέμονται στη ζωή του. Και φυσικά όλα αυτά δεν μπορούν να αξιολογηθούν χωρί να λάβουμε υπόψη κατά πόσον είναι βιώσιμα στο χρόνο και κατά πόσον ε, μπορούμε να έχουμε ευημερία για τι μελλοντικέ γενναίε. Δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή μία μέτρηση μια στιγμία εικόνα. Πρέπει να μετρήσουμε κάτι το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και τι μελλοντικέ καταστάσει. Είτε πρόκειται για ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, είτε για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Πρέπει να δούμε και τι γίνεται για τα εισοδήματα. Μιλάμε για αξιοπρεπεί μισθού, για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και αυτά έχουν σημασία. Και φυσικά ε, η καταλληλότητα των ε, κοινωνικών συστημάτων ασφαλείας. Επίσης θα πρέπει να προσμετρήσουμε και την ε, ε, αμοιβόμενη εργασία αλλά και την θελοντική εργασία, ε, δουλειά η οποία είναι αόρατη ορισμένες φορές αλλά συνεισφέρει τα μάλα στη συνοχή της κοινωνίας μας. Και τέλος, υπάρχουν μια σειρά από δείκτες πέραν του ΑΕΠ. Έχει, γίνεται πάρα πολλή δουλειά. Υπάρχει ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης. Η Eurostat έχει ένα δίκτυο ο οποίος λέγεται SALY και αφορά την ικανοποίηση και σε συνδυασμό με το προσδόκιμο ζωής. Μία τελευταία παρατήρηση, γιατί ξέρω ότι έχουμε να ψηφίσουμε στις 9.30 και θα ήθελα να δώσω χρόνο και στους συναδέλφους να κάνουν παρατηρήσεις, είναι ότι το ΑΕΠ είναι το πιο προφανές ε, στοιχείο ε, και ε, κατά την άποψή μου διαμορφώνει και την πολιτική και θα πρέπει να το εξετάσουμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω από όσου συζητούν κατηδίαν να σταματήσουν τα πηγαδάκια ή να βγουν έξω από την αίθουσα. Να δώσω τώρα το λόγο σε όσους ζήτησαν να μιλήσουν. Ο κύριος Σωρή και μετά η κυρία Κίνγκα Κούρτς. Α, έχω εγώ Μιλάω εξ ονόματος ε, του Τόμας Ντόιτς, ο οποίος είναι ο εισηγητής ε, από πλευράς ε, του ΕΛΚ, σκιώδηση της, γιατί χρειάστηκε να μεταβεί στο Βουκουρέστι σήμερα το πρωί. Είναι σε μια αποστολή παρατήρησης εξ ονόματος της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό δεν μπορεί να παραστεί σήμερα. Ε, συνεργάστηκα με την κυρία Χάρκιν και μου ζήτησε να παρουσιάσω ένα νέο τμήμα που προτείνει ο ίδιος και νομίζω ότι έχει συζητηθεί ήδη με την κυρία Χάρκιν και αφορά με την, ε, στη συνεργασία ε, σε τοπικό επίπεδο δήμων ε, και εφαρμογή μέτρων αυτής της μερφές. Μετά από το Totally, ε, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μην φαίνεται τόσο στεναρό αυτό το στοιχείο εδώ. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι δεν είναι κατάλληλο το ΑΕΠ, Απλώ πρέπει να πούμε ότι χρησιμοποιείται ο μηχανισμός αυτός εδώ και χρόνια και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διάφορες τάσεις και εξελίξεις. Δεν θεωρούμε ότι το ΑΕΠ είναι ακατάλληλο στοιχείο, αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι μεν κατάλληλο, αλλά πρέπει να το εξετάζουμε από κοινού και με άλλα ε, στοιχεία. Γι' αυτό ε, θα θέλαμε να γίνει αυτή η προσθήκη εδώ. Κατά τα άλλα, να ευχαριστήσουμε την κυρία Χάρκιν. Ε, συμφωνούμε με το σχέδιο γνωμοδότησής της. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ εκ μέρους των σοσιαλιστών θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζουμε πλήρως την πρωτοβουλία αυτή και φυσικά υποστηρίζουμε την δουλειά που έκανε η κυρία Χάρκιν. Το, α, δεν λέμε ότι το έπινε κατάλληλο, αλλά φάνηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης επειδή είχαμε ακριβώς τα οικονομικά στοιχεία, ε, είχαμε τα οικονομικά μεν στοιχεία, αλλά δεν είχαμε τα κοινωνικά δεδομένα. Οπότε αυτό δίνει ένα λόγο παραπάνω για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επί του θέματος. Το ΑΕΠ δεν μπορεί να ε, υπολογίσει τη διανομή των ε, ε, μισθών, ούτε πώς φτάνουν τα επιδόματα στον καθένα πολίτη. Και αυτό είναι πραγματικότητα σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν λοιπόν σημαντικό να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει το να μετρήσουμε την ποιότητα ζωής, νομίζω ότι χρειαζόμαστε άλλους δείκτες. Μπορούμε να το δούμε μέσω τροπολογιών ίσως. Συνεκτικότητα στην κοινωνία, κοινωνική συνοχή, ε, συμπερίληψη στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, ε, προσδόκιμο ζωής. Επίσης και, αυτό είναι, και αυτός είναι ένας δείκτης σημαντικός, πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής υπηρεσίας, πολιτισμό, μεταφορές, επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα, πρόσβαση σε πληροφόρηση, αξιοπρεπής εργασία, απασχόληση, ξεκούραση, ε, προφανώς έλλειψη διακριτικής μεταχείρισης, διακρίσεων, το συζητήσαμε και χτες και τον τελευταίο μήνα πρόσβαση σε υγιές περιβάλλον, ε, στέγαση, καθαρό νερό, θέρμανση, ε, σύστημα ε, διαχείρισης απορριμμάτων, ποιότητα ζωής, πρόσβαση στις νομικές, στις νομικές υπηρεσίες κτλ. Ελπίζω λοιπόν ότι θα καταλήξουμε σε ένα πολύ δυνατό εργαλείο για να έχουμε ένα νέο τρόπο να μετρούμε την, το ΑΕΠ. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζιν Λάμπερτ και μετά η κυρία Φιγκερέιδο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ την εισηγήτρια. Θεωρώ ότι η γνωμοδότησή της επιτυγχάνει να περιλάβει πολλές πληροφορίες μέσα σε πολύ λίγο αριθμό λέξεων. Η ομάδα μας σίγουρα συμφωνεί με την κεντρική ιδέα. Πάντα θεωρούσαμε ότι το ΑΕΠ είναι ένα πολύ στεγνό μέτρο που μετρά μόνο την, ποιότητα και την ποσότητα και δεν μετρά την ποιότητα. Ε, αν ο βασικός στόχος είναι το 3% κάθε χρόνο, 3% ε, ανάπτυξης, τότε αυτό δεν λέει σίγουρα τίποτα για την ποιότητα της παραγωγής και αυτό νομίζω ότι δείχνει ότι ε, κατατρώγουμε τον πλανήτη πολύ πιο γρήγορα. Ε, είναι πολύ σημαντική λοιπόν η γνωμοδότηση αυτή γιατί η Κωνσταντίνα έχει χαμηλότερη ανάπτυξη από την Νιγηρία αλλά είναι ισότιμη ε, κοινωνία με την Νιγηρία. Υποστηρίζουμε λοιπόν την έκθεση. Προφανώς θα υπάρξουν και κάποιες τροπολογίες, θα υποβάλουμε. Ε, και θα ήθελα να τονίσω και κάτι σε ό,τι αφορά την ε, διάσταση των δύο φύλων και το πώς ε, βλέπουμε τους δείκτες. Επίσης, η δουλειά που πληρώνεται και οι θέσεις εργασίας που δεν έχουν οικονομικό αντίκρισμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς κρατάει την κοινωνία ενωμένη, πώς μπορούμε να επιτύχουμε κοινωνική συνοχή. Όσο, μπορέ, όσο πιο γρήγορα μπορέσουμε να απομακρυνθούμε από το στεγνό ΑΕΠ, τόσο καλύτερα νομίζω ότι θα είναι τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Φιγκερέιδο και μετά η κυρία Μωράν. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ νομίζω ότι η συνάδελφός μας έχει κάνει πραγματικά μια πολύ καλή δουλειά. Μία σελίδα έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, αλλά έχει καταφέρει να συμπεριλάβει πολύ σημαντικές ιδέες μέσα σε αυτή τη μία σελίδα. Ε, απομακρύνεται από, τον, από το στεγνό ΑΕΠ και περνά σε πιο ποιοτικού αλλά και περισσότερου ε, ποσοτικού δείκτε που μπορούν να αντικατοπτρίσουν καλύτερα την πραγματικότητα. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Γενικώ συμφωνώ με τις διάφορες πτυχέ που αναφέρονται και στην έκθεση και που ακούστηκαν από τους ε, συναδέλφους, ας πούμε, ναι, θα πρέπει να δούμε το, τη διάσταση των δύο φύλων, την ισότητα μεταξύ άντρων και γυναικών, ε, πολιτιστικές πτυχέ, απασχόληση, ε, εργασία έμισθη και άμισθη. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν και, άλλες, υπάρχουν και κάποιες πτυχές που δεν έχουν θυγεί ακόμη. Μία σημαντική που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας για το μέλλον είναι η δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών δεν είναι αρκετό να έχουμε απλώς καλύτερη ποιότητα ζωής. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα συμμετέχουν. Γιατί αυτοί, γιατί θα, και ότι θα υπάρχουν μάλλον οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορούν να συμμετέχουν. Είτε θα είναι αυτό στην, στην τοπική τους ζωή, στην τοπική τους κοινωνία, στην περιφερειακή κοινωνία, σε διάφορα επίπεδα αυτοδιοίκησης. Επίσης, θα μπορούσαν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συμμετοχή ε, των εργαζομένων είναι σημαντική στην διαχείριση των εταιριών στις οποίες δουλεύουν. Ε, αυτό μπορεί να γίνει και σε επίπεδο περιφέρειας, τοπικό και σε εθνικό επίπεδο προφανώς. Οι εκπρόσωποι των, ε, εργαζομένων, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συνήθως έχουν ελάχιστες δυνατότητες να ακουστεί η φωνή τους. Σε μια κοινωνία λοιπόν που θα μπορεί να ζήσει στο μέλλον, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η δημοκρατική συμμετοχή ε, και οι σχετιζόμενες με αυτήν αξίες είναι σημαντικές και θα πρέπει να τις ε, έχουμε πάντα υπόψη και αυτό αν μπορεί θα ήθελα να το συμπεριλάβει η εισηγήτρια στην έκθεσή της. Ευχαριστώ. Η κυρία Μωράν και μετά ο κύριος Πουπάκης. Χωρίς μικρόφωνο, ομιλήτρια. Euh, euh, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την κυρία Χάρκιν για την εξαιρετική δουλειά της. Πράγματι αντιμετωπίζουμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Το ΑΕΠ είναι μία σειρά από μέτρα τα οποία ήταν χρήσιμα πριν από 50-60 χρόνια αλλά σήμερα πλέον πρέπει οπωσδήποτε να εξελιχθούν. Δεν βρισκόμαστε στην ε, ίδια περίοδο όπως, ήταν, ε, όπως βρισκόμασταν τότε που ασχοληθήκαμε με το δίκτυο του ΑΕΠ και το ακαθόριστο εγχώριο εισόδημα. Χρειαζόμαστε πλέον ένα στιγμιότυπο το οποίο μας επιτρέπει να δούμε τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή και να λάβουμε απόψη. Δεν θα ε, πρέπει να το βλούμε μόνο ως ε, την παρούσα κατάσταση, αλλά ως ένα μέσο το οποίο θα μας επιτρέπει να δούμε πώς πρέπει να διαμορφώσουμε τις πολιτικές μας. Ε, Όλα τα στοιχεία λοιπόν τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο δίκτυο του ΑΕΠ όπως ισχύει αυτή τη στιγμή πρέπει να εξελιχθούν και να συμπεριληφθούν κάποιο τρόπο. Και μεταξύ των νέων δικτών ε, υπάρχουν όλοι αυτοί που αναφέρατε που είναι πολύ σημαντικοί αλλά εγώ θα ήθελα να βρίσκονται και όλα όσα γίνονται σε κάθε χώρα για τη διαβίου κατάρτιση, όπου όπως έλεγε η κυρία Φιγκερέιντο πριν από λίγο, είναι το στοιχείο στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε απαραίτητο ε, προκειμένου να αναπτύξουμε το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή την αξία του εργαζομένου και που έχει να αλλάξει ε, τα επαγγελματικό του προσόντα για να μπορέσει να εξελιχθεί επαγγελματικά. Ε, το είδαμε και στις επιχειρήσεις στην Ιρλανδία η κυρία Χάρκιν ε, ξέρει πολύ καλύτερα από μένα ότι οι εργαζόμενοι σε μεγάλες επιχειρήσεις δεν είχαν καταρτιστεί ή επιμορφωθεί για τίποτα και φυσικά ήταν πολύ μεγάλο το βάρος της αλλαγής επαγγέλματος στη συνέχεια. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να επιμείνουμε σε αυτό και επίσης να επιμείνουμε και στην έρευνα, διότι η έρευνα είναι το μέλλον, οι δυνατότητες ανάπτυξης των επιχειρήσεων και βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο πνεύμα του να είναι τα πράγματα δυναμικά και να ρέουν και φυσικά ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την εθελοντική εργασία, συμφωνώ απολύτως. Ε, επίσης την ανάγκη να μετρήσουμε τις πραγματικές αξίες των μισθών, διότι όλοι αυτοί με τα τρίκουμπα κουστούμια θα σας πούνε ότι οι μισθοί είναι η τάδε, αλλά στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν είναι έτσι. Αυτά πρέπει να τα προσμετρήσουμε και επίσης πρέπει να δούμε και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν να συμφιλιώσουμε την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή, διότι δεν μπορεί να λέμε ότι έχουμε αξιόπιστο ΑΕΠ αν δεν έχουμε και αυτούς τους δείκτες. Τέλος, θα ήθελα να συμφωνήσω με ε, το συνάδελφο που είπε ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε το ΑΕΠ όχι μόνο ως στοιχείο εθνικής ε, κατεύθυνσης, αλλά θα πρέπει να το δούμε και σε περιφερειακό επίπεδο. Ε, πλέον σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές χώρες, στις οποίες υπάρχουν ε, οικονομικές ευθύνες στις περιφέρειες που είναι πάρα πολύ σημαντικές και δεν θα μπορέσουμε να έχουμε εθνικές κατευθυντήριες γραμμές αν δεν μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη και το περιφερειακό επίπεδο σε όλες αυτές τις κατευθύνσεις μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πουπάκης με τρίκουμπο κουστούμι. Ευχαριστώ. Φυσικά το ΑΕΠ δεν είναι ένα κατάλληλο στοιχείο. Ο κόσμο όμω δεν ζει μόνο με ΑΕΠ, μόνο με αριθμού. Πρέπει να βλέπουμε και τον άνθρωπο. Να έχουμε στο κέντρο την επιβίωση του ανθρώπου. Γιατί γι' αυτό ίσω χρειάζονται και άλλοι δείχτε. πολύ καλή η σύγηση, η τοποθέτηση, με ιδιαιτερότητε ίσω σε κάθε χώρο, χώρα, ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκεται η κάθε χώρα. Αυτό ήταν άλλωστε και το σύνθημα και τα αιτήματα οι ανησυχίε 50 ευρωπαϊκών συνδικάτων χθε που διαδήλωσαν, όπου και εγώ ήμουν παρόν, λέγοντα ο κόσμο όχι στι πολιτικέ λιτότητε για, την αντιμετώπιση τη κρίση, οδηγώντα τη φτώχεια, αλλά και ταυτόχρονα ζητώντα στήριξη στην ανάπτυξη και απασχόληση. Γι' αυτό ίσω, συμφωνώ και με τον κύριο Μαν, θα πρέπει να λάβει πρωτοβουλία στο τμήμα μα για αυτή, στην κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Νομίζω ότι αυτό το θέμα των δικτών ε, είναι ένα θέμα που το συζητούμε εδώ και καιρό σε σχέση με το ΕΠ. Και υπάρχει λόγος που πρέπει να συνεχίσουμε να το συζητούμε και ο λόγος αυτός είναι η κρίση την οποία βιώνουμε. Είμαστε στην ε, δεύτερη φάση αυτή τη στιγμή όπου μπορούμε να δείξουμε λίγη περισσότερη ευελιξία. Νομίζω όμως ότι πρέπει να πούμε γιατί η κρίση είναι ένας ε, λόγος που μας οδηγεί στο να επιλέξουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε κάποιες μακροπρόθεσμες ε, απόψεις οι οποίες ίσως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες τις οποίες όμως δεν θα γνωρίζουμε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα διοργανώνει, ε, εκπονεί την ε, στρατηγική της ε, για το 2020. Μπορεί να μα αρέσει, μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά αυτό είναι ο δικό μα χάρτης. Ο οποίος θα μείνει κενός νοήματος εάν δεν βασιστεί σε, κάποιες παραδοσιακές, σε κάποια παραδοσιακά κριτήρια του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ε, Έχουμε και την ε, Επιτροπή για την Οικονομική Κρίση, αλλά ελπίζω ότι μπορούμε και εμείς εδώ, στην, ε, μέσω της δικής μας Επιτροπής, να ξανακάνουμε την σύσταση προς την Κομισιόν. Να ξαναζητήσουμε δηλαδή από την Κομισιόν να αρχίσει να χρησιμοποιεί τους νέους δείκτες συγχρόνως με τους παραδοσιακούς δείκτες που χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια σύγκληση μεταξύ των δικτών που χρησιμοποιούμε. Στην παράγραφο 6 νομίζω ότι τα λέγονται είναι σημαντικά. Αλλά μιλούμε και για την ποιότητα της στέγασης. Για να είμαστε λοιπόν συνεπείς, θα πρέπει να μιλήσουμε και για την ποιότητα μεταφορών. Γιατί νομίζω ότι με τα στα εναλλακτικά κριτήρια οι μεταφορές, ο τομέας των μεταφορών είναι ένας τομέας ο οποίος αυξάνει το ΑΕΠ και βελτιώνει την ποιότητα ζωή των ανθρώπων με πολλού τρόπου. Επίση, πρέπει να μιλήσουμε και για την ποιότητα τη εκπαίδευση. Υπάρχουν λοιπόν κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν εδώ στην έκθεση. Ο δυναμισμό επίση που δημιουργείται μέσω τη κοινοτομία και όλα όσα συνδέονται με αυτό. Κυρία Χάρκιν, στην παράγραφο 2 ασχοληθήκατε με το θέμα αυτό και με την ανάγκη να εμπλακεί περισσότερο, να συμμετάσχει περισσότερο η κοινωνία σε μια κοινή στρατηγική και την δυνατότητα που έχει η κοινωνία να είναι καινοτόμο. Πιστεύω ότι η δυνατότητα για καινοτομία δεν καλύπτεται από τους ε, παραδοσιακούς δείκτες για το ΑΕΠ. Νομίζω λοιπόν ότι στην αγρονομοδότηση που θα δώσουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα πρέπει να αναφέρουμε και το ρόλο που παίζουν οι, οι δημόσιες υπηρεσίες στην ποιότητα ζωή, ζωής των πολιτών και θα πρέπει να μετρήσουμε την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών που παρέχονται. Αυτά είναι τα δικά μου σχόλια για να συμπληρώσω την εξαιρετική σας κατά τα λοιπά ε, γνωμοδότηση. Δεν ξέρω κυρία Χάρκιν αν θέλετε να πάρετε το λόγο για να κάνετε κάποια τελειωτικά σχόλια. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη γιατί ξέρω ότι θα πάμε και στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, εξαιρετικές οι ιδέες τους, καινούριε οι ιδέες τους, οπότε φαίνεται ότι έχω και άλλη δουλειά και πραγματικά προσβλέπω στην καλή μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Euh, nous allons donc ouvrir un délai dépôt des amendements. Ευχαριστώ. Προθεσμία κατάσταση τροπολογιών 12 Οκτωβρίου το μεσημέρι και θα τις εξετάσουμε στα μέσα Νοεμβρίου για να τα εγκρίνουμε αργότερα στην Ολομέλεια και ε, η Επιτροπή Περιβάλλοντος που είναι επί της ουσίας Επιτροπή λογικά θα ε, πρέπει να αποφασίσει στις 29 Νοεμβρίου ή στην 1η Δεκεμβρίου. Να περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Ελπίζω να έχετε όλες τις κάρτες σας. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει έρθει χωρίς κάρτα. Ο κύριος Ορή. Στην προηγούμενη συνεδρίαση των συντονιστών δεν ήταν σαφές τι θα γίνει με την έκθεση για τους Ρωμά. Η πρόεδρος έλαβε μια απόφαση με την οποία εγώ διαφωνώ και εγώ θα ήθελα να την ψηφίσουμε αυτή την απόφαση στην Επιτροπή. Ο κύριος Θέρκας. Κυρία Πρόεδρε, Ή εγώ δεν ήμουν στην ίδια συνεδρίαση με τον κύριο Ρή, ή δεν ήταν σαφές ότι η έκθεση για τους Ρωμαί και η γνωμοδότηση που θα πρέπει να ετοιμάσει η Επιτροπή μας για την Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων ήταν έκθεση που θα πρέπει να αναλάβουν οι σοσιαλιστές. Οι σοσιαλιστές τη ζήτησε γιατί το ΕΛΚ δεν ήθελε να κάνει έκθεση για το θέμα. Και επειδή την ε, επί της ουσίας έκθεση θα κάνει από την Επιτροπή Πολιτικών ε, Ελευθεριών ε, το ΕΛΚ ζητήσαμε εμείς τη γνωμοδότηση να την κάνουμε εδώ στους σοσιαλιστές. Δεν καταλαβαίνω κυρία Πρόεδρε γιατί θα πρέπει να συζητηθεί στην Επιτροπή και να ψηφίσουμε ένα θέμα το οποίο ήταν σαφέστατο στους συντονιστές. Έχουμε βέβαια και τους άλλους συντονιστές εδώ οι οποίοι μπορούν να επιβεβαιώσουν αυτό που μόλις σας είπα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Θέρκας. Συμφωνώ. Τα πρακτικά της συνεδρίασης των συντονιστών ε, λένε αυτό που λέτε κι εσείς. Δεν υπήρξε κανένας δισταγμός για την απόφαση που ελήφθησε στην ε, συνεδρίαση. Να περάσουμε λοιπόν στο σημείο 7. Η δημογραφική πρόκληση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Έκθεση του κυρίου Τόμας Μαν. Έχουμε και δύο γνωμοδοτήσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Γυναικών. Και παρουσιάστηκαν τροπολογίες ε, για την ε, παράγραφο 1. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μετά από την παράγραφο 1 Παράγραφος 32 με τροπολογία του κ. Χίγγινς Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 2. Συμβασμός D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Κυρία Τζίμερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 3, συμβιβαστική τροπολογία ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 4, συμβιβαστική τροπολογία F, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία G, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά, ένα Επιτροπή Γυναικών, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53. Καμπνόχ υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές σε ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ναι, ναι, ψηφίσατε. Πέρασε ψηφοφορίας. ψηφοφορία έχει πρόβλημα. Δεν ξέρω, δοκιμάστε το άλλο μηχάνημα. Ορίστε, κανένα πρόβλημα. Ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας, 24 υπέρ, 19 κατά, εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία 54. Ροντζούλη Μπαλντασάρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55. Χάρκιν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56. Τζίμερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κατόπιν. Euh, Τροπολογία 57. Κοζά υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11. Επιτροπής Γυναικών υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 κάστεξ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική AX, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Γυναίκες 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 69 της κυρίας Λίν. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. 23 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται με μία αποχή. 70 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία I υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, 74, ε, τροπολογία διαγραφής από τον κύριο Καμπρινόχ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία J, λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Συμβαστική τροπολογία K. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ανεξάρτητα από τη συμβαστική τροπολογία ΚΕΙ, οι πράσινοι θέλουν να θεωρηθεί ως προστίκη το Life Cycle Approach to Employment Ωραία. Ε, μόλις ψηφίσαμε τη συμβαστική τροπολογία K, και θα ήθελα να ρωτήσω από τον συγητή και τους υπολείπους αν δέχονται μια προφορική τροπολογία για να αντικατασταθεί ο όρος flexicurity με το life cycle approach to employment. Κύριε συγητά. Ε, Συμφωνώ. Υπάρχουν ενστάσεις για την προφορική τροπολογία. Κύριε Έγγελ. Μήπως άπρεπε έπρεπε να καθόμαστε, να σκεφτόμαστε γενικότερα τι ακριβώς συμβαίνει, η flexicurity, δηλαδή και μετά το κάνουμε και life cycle approach. Τι είναι, μπαταρία ε, επαναφορτιζόμενη. Τέλος πάντων, η προφορική τροπολογία δεν γίνεται δεκτή, λέει η Πρόεδρος, και περνάμε λοιπόν στη τροπολογία 90 της κυρίας Κάστεξ, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία L, παράγραφος 13, με προφορική τροπολογία του εισηγητή και της ομάδας των σοσιαλιστών. Ποιος είναι υπέρ της συμβαστικής τροπολογίας L με την προφορική τροπολογία. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 94 της κυρίας Μπλινκεβιτσιούτη υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 96 με προφορική τροπολογία των φιλελευθέρων. Και νομίζω ότι τη δέχεται και ο εισηγητής. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 98 του κυρίου Πουπάκη υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 99 του ιδίου υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 10 Επιτροπής Γυναικών υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 100 της κυρίας Χάρκιν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 103 της κυρίας Όμεν Ρόιτε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 102 κόσα υπέρ, κατά κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική τροπολογία M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, έχετε δίκιο. Και πάλι στην παράγραφο 16, τροπολογία 116 της κυρίας Κορνέλισεν με προ... ε, έτοιμα για κατάτμήματα ε, ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα μέχρι το working trading, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το υπόλοιπο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 16. 117 της κυρίας Πλάμ με ε, κατά ψηφοφορία το πρώτο μέχρι το opportunity υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 Τζίμερ υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 119 από έτσι διαγραφής υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία N με προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ της N με την προφορική τροπολογία. Contre, Κατά, αποχές, εγκρίνεται. après le Κυρία Λίν, έχει ε, ζητήσει προσθήκη στην 120 το τμήμα της ε, τροπολογίας της που αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ε, μη διάκριση. Ποιοι είναι υπέρ της προσθήκης αυτής κατά, αποχές, απορρίπτεται. τον παράγραφος 17, ε, οι 124 και 125 που είναι ε, αιτήσει για διαγραφή. Κυρία Λάμπερτ. Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά αν δείτε την 120 ως προσθήκη, την ψηφίσαμε μεν, αλλά την 84 δεν την πήραμε σαν προσθήκη δεν είναι προφορική η τροπολογία, ήταν συγκεκριμένο κείμενο. Δεν, είναι, δεν υπάρχει μια συνέπεια εδώ. Μήπως πρέπει να ξαναδούμε την 84. Δεν είναι προφορική η τροπολογία 84, υπάρχει κείμενο. Και αφού το κάναμε για την ε, τροπολογία της κυρίας Λίνη το 120, το κάνουμε και για την 84. Δεν θα ξεκινήσουμε συζήτηση τώρα. Το θέμα είναι σαφές. Ε, είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο απορρίφθηκε αυτή η τροπολογία. Περνάμε λοιπόν στην παράγραφο 17 σημείο 2. Ε, οι 124 και 125 και 126 ζητούν διαγραφή. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 127 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 128 της κυρίας εν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 17 σημείο 2α. 129 της κυρίας Πλάμ με κατατμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα μέχρι το restructuring υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτό 130 της κυρίας Κορνέλησεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Σημείο 4. Δύο προπολογίε διαγραφή 132 και 133 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία ΟΟΥ υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στην 138 υπέρ. Κατά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 κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση για τη συμβιβαστική τροπολογία Β. Tout le monde a pu voter? Ψήφισαν όλοι. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 15 υπέρ, 28 κατά, είχατε απόλυτο δίκιο. Δεν εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία Β, επομένω ψηφίζουμε την 159 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 155 είναι συμβατή από τη φαίνεται υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 157 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κατόπιν 160 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 161 υπέρ ε, κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία Q υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 167 παράγραφος 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε την 166. Tout le monde a pu voter. Ψήφισαν όλοι πέρασε της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 19 κατά. Έχετε δίκιο, εγκρίνεται. 164 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 165 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία R, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 172 κάστεξ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 173 αποπάκης υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 174 ράπτη υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται. 175 υπότιτλος 10 υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. Παράγραφος 24. Συμβιβαστική τροπολογία S ε, βάσει του κειμένου που σας έχει διανεμηθεί, το οποίο ε, τροποποιήθηκε. Θέλετε να σας διαβάσω την τελική εκδοχή ή ε, τους εμπιστεύεστε, τους συντάκτες. Ωραία, ψηφίζουμε υπέρ. Κατά, δεν είναι τόσο βέβαιο για να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 16 υπέρ, 27 κατά. Απορρίπτεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 180 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 177 κορνελίσαν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 176 είναι συμβατή, υπέρ, συγγνώμη, καταπίπτει 176, μπορούμε να ψηφίσουμε όμως την 178 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι πέρας, 22 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται. 181 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Γυναίκες 6 υπέρ, κατά αποχές να ευαληθεύσουμε για την έξι είναι πολύ πιο σαφές τώρα ψήφισαν όλοι πέρασε ψηφοφορίας 30 υπέρ 9 κατά εγκρίνεται 182 Βλικιβιτσιούτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25. 183 του κυρίου Τσάμπνοχ υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ταφ. Α, να το ελέγξουμε. Ωραία, να ελέγξουμε την 183. Tout le monde a pu voter. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε φορέας. 11 υπέρ, 31 ψήφι κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική ταφ υπέρ. Κατά. Απόχες. Έγκρινεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 126. Ε, παράγραφος 26, συγγνώμη, 192. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 189. Υπέρ κατά αποχε εγκρίνεται 190 πουπάκης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 191 Jim Higgins υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 Μπαχ υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται γυναίκες 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, ε, πέντε των γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 παράγραφος ακόμα 194 λίν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 197 195 συγγνώμη κυρία Πλικεβιτσούτε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 198 λιν 20, ε, παράγραφος 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 199 κόζα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Αν να το ελέγξουμε. Αν θέλετε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 200. Ε, Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 22 υπέρ, 18 κατά. Μία αποχή εγκρίνεται. 201, M. Kozak, που. 200 του κυρίου Κόζα. 201. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 202. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 203. Υπέρ. Κατά. Ποιος είναι υπέρ για την 203. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 205. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. «204 καταπίπτει». Πάμε στην 206. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 207. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 208. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 209 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά Tout le monde a pu voter Le vote est clos. 21 ψήφοι υπέρ, 20 κατά εγκρίνεται. Πάμε στην παράγραφο 30. Πάμε στην μητρία των γυναικών, συγγνώμη. Υπέρ, κατά, αποχές, 13, ε, εγκρίνεται. 13 των γυναικών, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.14, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 215, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 216 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 217 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 218 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 219 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 τροπολογία 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 221 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 222 υπέρ κατά να το ελέγξουμε ελέγχουμε τη 222 Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Πέρας ψηφοφορίας, 22 ψήφοι υπέρ, 17 ψήφοι κατά, εγκρίνεται. 2.23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.24 να το ελέγξουμε να ελέγξουμε την 2.23 Tout le monde a pu le vote Πέρας 24 ψήφοι υπέρ, 18 ψήφοι κατά. Είχατε δίκιο. Εγκρίνεται. 2.24. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 32, τροπολογία 225. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 228. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 226. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.27 είναι συμβατή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 2.29 Πουπάκης. Υπέρ. Κατά. Κατά, Εγκρίνεται. 2.30 υπέρ. Κατά. αποχε Εγκρίνεται. 2.31 υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 2.32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.33 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 14 των γυναικών, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.34, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.35, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.36, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.37, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.38 Χίρς με τροπολογία προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.39 παράγραφος 34 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε ελέγχουμε τη 2.39 Tout le monde le 23 ψήφοι υπέρ, 18 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. 2.40 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.42 ηλίν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.43 παράγραφος 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.46 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές να ελέγξουμε τη 2.46 Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Πέρας ψηφοφορίας. 25 ψήφοι υπέρ, 17 κατά εγκρίνεται. 2.47 που πάκης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παράγραφ 4 de la Commission des Femmes qui pour. 4 των 4 γυναικών υπέρ κατά εγκρίνεται. 2.49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.50. Τόμας Μάν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε. Πάμε στο 1. Λιν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται 14 κάστεξ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος β των γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σ των γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική Β. Υπέρ. Συμφωνείτε να προσθέσουμε στη συμβαστική B την τροπολογία 19 της κυρίας Λίν. Όχι. Ναι, αλλά δεν έχει συμφωνηθεί ω ε, προφορική τροπολογία. Είναι προσθήκη. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ήδη το έχουμε κάνει δύο φορέ. Δεν θα αλλάξουμε τώρα του κανόνε. Λοιπόν, συμβαστική Β. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Ναι, αλλά αν υπάρχει συμβαστική πρόταση για μια παράγραφο και ο εισηγητή και ο συντάκτη τη της παραγράφου θεωρεί ότι μπορεί να καλύψει κάποια τροπολογία, δεν μπορούμε να μετανορθούμε και να πούμε είναι προσθήκη ο εισηγητής θεωρεί ότι καλύπτεται. Είναι τριών ε, εισηγητών, είναι τριών εισηγητών η τροπολογία, λέει η κυρία Λίν, ο κύριος Μαν. Λοιπόν, η συμβαστική Β ε, ψηφίστηκε και εγώ θα καταψήφιζα την κυρία τη 19 και ως προσθήκη και ως οτιδήποτε θα την καταψήφιζα. Οπότε η τροπολογία της κυρίας Λίν δεν καλύπτεται, λέτε, από τη συμβαστική τροπολογία. Αυτό εννοείται. Ε, ίσως, για να μην έχουμε προβλήματα διαδικαστικά, ας ψηφίσουμε κανονικά και για τα δύο. Και για την τροπολογία της κυρίας Λίν. Νομίζω ότι είναι πιο δίκαιο αυτό. Λοιπόν, ψηφίζουμε τη 19. Αν είναι προφορική τροπολογία, εγώ είμαι αντίθετη. Δεν είναι προφορική τροπολογία, δεν καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία, οπότε θα την ψηφίσουμε κανονικά. Πάμε στη 19 της κυρίας Λίν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Οπότε να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Sur Ψηφίζουμε την τροπολογία της κυρίας Λίν. 19. Tout le monde a pu voter, le vote Πέρας ψηφορίας. 20 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην αιτιολογική δέλτα. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 24 Τόμας Μάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε να ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Tout le monde a le vote est clos. Πέρας ψηφοφορίας. 38 υπέρ, 2 ψήφοι κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Να πάμε τώρα στην ε, γνωμοδότηση του κ. Νταβίτ Κάσα για την βελτίωση τη οικονομική διακυβέρνηση και του πλαισίου σταθερότητα τη Ένωση, ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ. Παράγραφο 1, τροπολογία 6. Υπέρ.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 Après Περνάμε στην τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18. Συμβατή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20. Του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ της κυρίας Γκρουνή η τροπολογία που θα πρέπει να θεωρηθεί ως προσθήκη αυτό μου γράφουν εδώ 22 λοιπόν ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 του κυρίου Κοφεράτη υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Την 23 ελέγχουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέραση ψηφοφορία. 16 υπέρ, 24 κατά. Είχατε δίκιο, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 24 του κυρίου Πιπάκη. υπέρ. Κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 25 παράγραφος 6. Του κυρίου Κοφερά... Ο κύριος Κοφεράτη ζητάει το λόγο. Αποσύρω την τροπολογία 25. Μπορεί να την ξαναπαρουσιάσω αργότερα. 25 αποσύρεται λοιπόν. 26 που και υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6, 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, ε, συμβαστική τροπολογία β υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στον υπότιτλο και την παράγραφο 7, α νέα, μετά από την 7, υπέρ, τροπολογία 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 8, 36, ε, διαγραφή υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 38 είναι συμβατή, ε, ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 ως προσθήκη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Υπότιτλος ε, και μια νέα παραγραφός μετά από την 8, η 40 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1 εισηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται ε, σκέψη α του Καφεράτη υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη β, 3 του ιδίου υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη β, 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε λοιπόν το σύνολο της γνωμοδότησης ε, ηλεκτρονικός άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 35 υπέρ, 6 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ελπίζω η γνωμοδότηση αυτή να εμπνεύσει τους συναδέλφους της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής, ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ομάδα Εργασίας του κ. Φαν Να περάσουμε τώρα στην... στην κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμοποίηση και να ψηφίσουμε κατά σειρά τις τέσσερις επιστολές για την ε, συνάδελφό μας την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε και τις τέσσερις μαζί. Εξαιρετικά. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Nous devons encore και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Λάμπερτ για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού 883 του 2004 και του κανονισμού δεν ξέρω ποιο ε, για του υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τι εν λόγω διατάξεις μόνο λόγω της ηθαγένειά τους. Και πριν ψηφίσουμε θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Λάμπερτ. Όχι, δεν θέλετε. Ωραία. Ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Η έκθεση της κυρίας Λάμπερτ εγκρίνεται ομόφωνα. Συγχαρητήρια κύριε Λάμπερτ. Δεν μας μένει λοιπόν παρά να εγκρίνουμε το σχέδιο χρονοδιαγράμματος των συνεδριάσεων της Επιτροπής μας για το 2011. Είναι κάποιος αντίθετος στο πρόγραμμά μας? Δεν είναι. Ωραία. Εγκρίνεται το χρονοδιάγραμμα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία και να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Τζίμερ για την παρουσίαση της γνωμοδότησής της για την έκθεση της Επιτροπής Γυναικών για το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Τζίμερ, έχετε... <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. για την ε, γνωμοδότηση και το, γυναικείο, το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρώπη. Μιλούμε για μια γνωμοδότηση που θέλει να ενισχύσει την ε, συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με την Επιτροπή ε, των Γυναικών. Γι' αυτό θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή, γιατί εδώ υπάρχουν ιδιαίτερες ρυθμίσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι λέω. Ωραία. Από την άποψη της Επιτροπής Απασχόλησης, εμείς με τη δική μας νομοδότηση, εάν τελικά ψηφιστεί όπως έχει στην Επιτροπή μας, θέλουμε να ε, προωθήσουμε κάποιες διατυπώσεις οι οποίες ε, στην, ε, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην γνωμοδότηση της Επιτροπής των Γυναικών. Οπότε εμείς ως Επιτροπή Απασχόλησης πρέπει να δείξουμε κυρίως την πτυχή των κοινωνικών διαστάσεων και με αυτή την βάση κάνουμε τις προτάσεις μας. Ε, οι οι απαιτήσει από την Επιτροπή Γυναικών θα πρέπει να παραμείνουν, ε, ή καθ' αυτού ε, προτάσει για τι γυναίκε θα πρέπει να παραμείνουν στην Επιτροπή Γυναικών. Η Επιτροπή Γυναικών, στα πλαίσια αυτή τη εκθέσεω, έχει οργανώσει μία ακρόαση, στην οποία έλαβα και εγώ μέρο και είχα την δυνατότητα και ω εισηγήτρια να μιλήσω για την γνωμοδότησή μου και ε, ε, αισθάνομαι ενισχυμένη γιατί αυτό το οποίο επέλεξα, ο τρόπος με τον οποίο επέλεξα να προχωρήσουμε είναι σωστός. Δηλαδή έχω συντάξει μια γνωμοδότηση η οποία δεν ε, έχει συγκεκριμένη, δεν περιλαμβάνει κάποιο συγκεκριμένο, κάποια συγκεκριμένη πτυχή των, της κατάστασης των γυναικών, είναι γενική. Γιατί και από την Επιτροπή Γυναικών δεν υπάρχει σχέδιο ε, γνωμοδότησης. Μιλάμε δηλαδή για συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες να προκύπτουν από την ε, ε, Επιτροπή των Γυναικών ε, και κάποιες που δεν έχουν συμπεριληφθεί από την Επιτροπή των Γυναικών εμείς μπορούμε με κάποιες τροπολογίες να τις συμπεριλάβουμε στη δική μας νομοδότηση. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι σκόπιμο να γίνει και στη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε. Να προτείνουμε δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα, να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι θα μπορούν ε, να βρουν ένα πλαίσιο στην ε, έκθεση που προετοιμάζει η Επιτροπή Γυναικών, συμπεριλαμβάνοντας πτυχές κοινωνικές, οικονομικές και προβλήματα των γυναικών. Πρώτον, ως Επιτροπή θα πρέπει να καταδείξουμε ότι και μετά την ε, οικονομική κρίση πλήττονται και η οικονομία και η κοινωνική η ανεργία στις, ε, στα κράτη-μέλη και γι' αυτό ζητείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει. Αυτή είναι μια συζήτηση που την κάνουμε σταθερά. Πρέπει να δεσμευθεί ώστε να, παρα... να απαλείψει τη φτώχεια και κυρίως τη φτώχεια των παιδιών. Μιλούμε για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φτώχειας και ε, κοινωνικού αποκλεισμού. Έχοντα λοιπόν υπόψη αυτό και ότι εμείς ως είμαστε Επιτροπή απασχόληση εμπλεκόμαστε στην όλη διαδικασία εκπόνησης ή συζήτηση του Μελλοντικού Ευρωπαϊκού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου το οποίο επίσης θα πρέπει να έχει ε, ακριβώς αυτό ως στόχο και εγώ έχω αναλάβει να αναφέρουμε και, την, ε, και, μια, και κάποια στοιχεία για τα οικονομικά ε, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να υπάρξουν δηλαδή μέτρα για, ε, κονδύλια συγγνώμη, για μέτρα, για δράσεις, για την στρατηγική, για την, προς, για την πρόθεση της κοινωνικής ένταξης και με βάση την πρωτοβουλία που υπάρχει για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Και αυτό θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια της Στρατηγικής Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Μεταξύ άλλων, να πω ότι Αυτή την ειδική πτυχή που την συζητήσαμε θέλαμε να την συμπεριλάβουμε και στο κείμενο. Ότι δηλαδή το θέμα των δικτών της φτώχειας είναι ουσιαστική βάση ώστε ακριβώς και λόγω της φτώχειας των γυναικών να έχουμε την ε, κατάλληλη βάση ώστε να έχουμε συγκρίσιμα δεδομένα και σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της κατάστασης και την εκπόνηση μέτρων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι δείκτες φτώχειας, έτσι όπως τους έχει ορίσει εκ νέου το, το Συμβουλίο, τους έχει διευρύνει εν πάση με τον καθορισμό του ότι τα κράτη-μέλη από την πλευρά τους θα πρέπει να επιλέξουν από μόνα τους τους ε, δείκτες που τους ταιριάζουν περισσότερο, θεωρώ ότι είναι ένα σημείο το οποίο ε, πρέπει να έχει δική θέση στην όλη συζήτηση για τη φτώχεια και κυρίως για τη φτώχεια των γυναικών. Έτσι όπως έζησα εγώ τη συζήτηση στην Επιτροπή των Γυναικών δεν έγινε αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε. Και επίσης μιλούμε για το πρόβλημα της κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής πολιτικής, και μιλούμε για την αναγκαιότητα μεμονωμένων νομικών απαιτήσεων, που, δικαιωμάτων που έχουν, τα, που έχουν οι γυναίκες ε, από τα κοινωνικά συστήματα. Από, με, από κοινού λοιπόν με την Επιτροπή Γυναικών νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια αρκετά ισχυρή έκθεση που να μπορεί να ψηφιστεί, να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο. Πρέπει να πω ότι είχαμε τέτοιε τέτοιες και στην τελευταία θητεία, στην προηγούμενη θητεία, γιατί εμείς ως Επιτροπή Απασχόλησης ήμασταν η καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή για την, ε, για την γνωμοδότηση και την αντιμετώπιση της φτώχειας του κοινωνικού αποκλεισμού και κυρίως της φτώχειας των παιδιών. Και πάλι η Επιτροπή των Γυναικών είχε τον ρόλο του να συνεργαστεί πιο στενά μαζί μας έτσι ώστε να καταφέρουμε με ένα συγκρίσιμο τρόπο να δράσουμε. Και το κάναμε και θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή και εκείνη η γνωμοδότησή μας και είχαμε λάβει μεγάλη πλειοψηφία. Αυτά από μένα, Πρόεδρε, για την πρώτη αυτή φάση, για την υποβολή του σχεδίου. Ε, κατά τα Μπορούμε να συζητήσουμε και για τροπολογίε. θα δούμε τι θα γίνει και με τις προτάσει των συναδέλφων και να δούμε με, από κοινού με την ε, Επιτροπή των Γυναικών πώς μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα πιο συγκεκριμένα. Bien, merci beaucoup. Ε, ωραία, ευχαριστώ. Oui. Euh... Madame Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τζίμερ, ε, συντάκτρια της νομοδότηση. η οποία μας είπε ποιες είναι οι πτυχές τις οποίες θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και εμείς στην έκθεση της Επιτροπής Γυναικών ε, μέσω τροπολογιών. Θα πρέπει λοιπόν καταρχάς να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε γενικές γραμμές ως προσθήκη και τι θα ετοιμάσει, σε αυτά που θα ετοιμάσει η Επιτροπή Γυναικών. Θα ήθελα να πω ότι η ανεργία, κυρίως η γυναική ανεργία θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια και αυτό δείχνει λίγο πολύ και την ε, ανεργία των ε, γυναικών τη φτώχεια μάλλον των γυναικών. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή ζωή και ε, να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις γυναίκες προσφέροντά του μια θέση εργασία. Πρέ, πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν κατάλληλα κίνητρα ώστε να δημιουργήσουμε απασχόληση και θέσει εργασία. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο σημείο, σίγουρα θα πρέπει να αυξήσουμε τις ε, χρηματοδοτήσεις, ε, διότι νομίζω ότι είναι ελλειπής αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να καταλάβουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με πιο καλά στοχευμένο τρόπο τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας. Σαφώς η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 περιλαμβάνει και την καταπολέμηση της ένδυας και του κοινωνικού αποκλεισμού και εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις πτυχές. Όμως είναι πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα της συγχρηματοδότησης για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Ακόμα συζητάμε πώς ε, θα μπορέσουμε να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συγχρηματοδότηση για την καταπολέμηση της γυναικείας φτώχειας και της παιδικής φτώχειας. Ε, ε, και εκεί υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε περιβάλλον απόλυτης ένδυας ε, και η οικογένειά τους δεν έχει ε, άτομα που να απασχολούνται σε καμία θέση εργασίας. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το συμπεριλάβουμε λοιπόν και αυτό στην έκθεση γιατί πάρα πολλά παιδιά που βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ αρνητικό στοιχείο. Ε, όπως έλεγε η κυρία Τσίμερ ε, στο σημείο 4, ίσως τα κράτη-μέλη δεν δρούν όπως θα έπρεπε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη μέρημνα για, το, ε, για την αρχή της επικουρικότητας, να βλέπουμε τι κάτουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη ε, για την συστηματική καταπολέμηση της φτώχειας και πώς προσπαθούν να καταπολεμήσουν τη γυναικεία φτώχεια αλλά στην προσπάθεια καταπολέμησης της φτώχειας υπάρχουν και κάποιες πτυχές οι οποίες είναι αλληλένδετες. Η υγεία, η απασχόληση, η παιδεία και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και η χρήση των βέλτιστων πρακτικών. Η κοινωνική προστασία αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της κοινωνικής ένταξης για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα της παιδείας, στον τομέα της επιμόρφωσης ε, και της απασχόλησης. Μας ε, ενδιαφέρει και το θέμα πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το πώς φτάνει κάποιο στο χώρο της εργασίας του. Ε, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία επιτρέπουν να ξεφύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο τη φτώχεια. Σε γενικές γραμμές ε, συμφωνώ, ε, θα παρουσιάσω μόνο κάποιες τροπολογίες ε, για τα σημεία στα οποία δεν συμφωνώ απολύτω και στη συνέχεια θα γίνει φυσικά συζήτηση επί των τροπολογιών. Η κυρία Πλάν και στη συνέχεια η κυρία Μωρά. Καλημέρα ε, σε όλους τους συναδέλφους και ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις τους. Εγώ είμαι η συγγήτρια στην Επιτροπή Γυναικών επί του θέματος. Η έκθεση δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένη, ε, είμαστε ακόμα επί το έργων, έχουμε μια πρώτη ε, προθεσμία στις 8 Νοεμβρίου. Ε, μελετήσαμε το σχέδιο κειμένου που έχει παρουσιάσει η κυρία Τσίμερ, θα το εξετάσουμε και επειδή έχω συνεργαστεί πάρα πολύ καλά με την Επιτροπή Απασχόλησης στο παρελθόν και με τα μέλη της Επιτροπής, έγινε και μία ε, δημόσια κρόαση πάρα πολύ καλή επί του θέματος Ε, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία λάβαμε από αυτή την ακρόαση και θα συμπεριλάβουμε στην ε, έκθεση. Ξέρουμε ότι η γυναική αυτόχεια έχει τρεις διαστάσεις. Τη, διάσταση του φύλου, τη διάσταση τη γεωγραφική και τη διάσταση των γενεών. και θα πρέπει να δούμε και τους στόχους που θέτει η στρατηγική της ε, Ευρώπης για το 2020 και το στόχο της μείωσης της ε, ένδυας και της ε, αύξησης της απασχόλησης και φυσικά τους στόχους της χιλιοκητίας και όλα όσα συνδέονται με την πορεία της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. η έκθεση θα περιλαμβάνει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της απασχόλησης των γυναικών, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, διακρίσεις στην αγορά εργασίας ε, για τις γυναίκες και θα πρέπει να αναφερθούμε στα αυτά τα στοιχεία διότι υπάρχει εδώ και η σχέση του pay gap, του χάσματος των μισθών ε, διότι υπάρχει και μία άμεση σχέση με ένα βιώσιμο σύστημα συντάξεων. Υπάρχουν κάποιες χώρες στις οποίες έχουν γίνει ίδιες μεταρρυθμίσεις ε, και θα πρέπει ε, να δούμε τι γίνεται εδώ και να λάβουμε υπόψη και το θέμα των συντάξεων γιατί έχει άμεση σχέση με το θέμα. και επίσης θα πρέπει να εντοπίσουμε και τα δικαιώματα που δίνονται από τα συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε στην ακρόαση και θα πρέπει να δημιουργήσουμε και θέματα κοινωνικής ένταξης για τις ε, γυναίκες μετανάστριες, για γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στις ευάλωτες ε, ομάδες, σε μειονότητες, διότι υπάρχουν προβλήματα ε, όπως για παράδειγμα με τους Ρωμά και φυσικά θα πρέπει να δώσουμε ε, μεγάλη έμφαση ε, σε θέματα συμφωλίωσης οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Αναφέρομαι σε όλα τα θέματα της ε, μητρότητας, των συνθήκων ασφαλείας και υγείας των γυναικών, καθώς επίσης και την άδεια μητρότητας. Ε, διαβίου μάθηση, ε, ε, νέες δεξιότητες για να μπορέσουν να είναι ενεργές στην αγορά εργασίας και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το, τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την βοήθεια των γυναικών και φυσικά προσβλέπω στην αγαστή συνεργασία για αυτή την έκθεση διότι πρόκειται για μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας και η οποία θα καταλήξει σε μέτρα με τα οποία μπορούμε ε, να κάνουμε κάποια πράγματα είτε σε νομοθετικό είτε σε νομιθετικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε πλέον συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα υπάρξει καλή συνεργασία με τους συναδέλφους και θα καταφέρουμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε ε, και ελπίζω στην ανοιχτή συνεργασία για να μπορέσουμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μωράν και στη συνέχεια η κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συναδέλφους, ε, την κυρία Τζίμερ και την κυρία Πλάμ για τις παρεμβάσεις τους. Θεωρώ ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών, την ισότητα μεταξύ των πολιτών, την καταπολέμηση της ένδυας και θα ήθελα να σταθώ λίγο στον ακριβή τίτλο αυτού του σχεδίου γνωμοδότησης. Το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φρονώ ότι ο κίνδυνος που ελεγχεύει εδώ είναι να προσπαθήσουμε να τα βάλουμε όλα σε μία τέτοια έκθεση. Να θα σας πω κυρία Τσίμερ ότι υπάρχουν πολλά σημεία στην ε, γνωμοδότησή σας ε, τα οποία με βρίσκουν απόλυτα συμφωνή, αλλά διαφωνώ σε ένα σημείο. Κάνετε μία ανάμιξη της ε, φτώχειας των γυναικών με τη φτώχεια των παιδιών, διότι για την παιδική φτώχεια έχουμε άλλους πόρους, άλλα προβλήματα και πρόκειται για ένα θέμα τελείως διαφορετικό το οποίο χρειάζεται τις δικές του απαντήσεις. Νομίζω ότι αποδονομώνουμε και τη δική μας την έκθεση για τη γυναική αυτόχεια, αλλά ε, ουσιαστικά χάνουμε και όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν και πρέπει να γίνουν για την ένδυα των παιδιών. Νομίζω λοιπόν ότι η παράγραφος ε, ε, που αφορά στην ε, παιδική φτώχεια, όπως είναι διατυπωμένη αυτή τη στιγμή, η παράγραφος 3, δεν είναι καλή και δεν μπορούμε να στόχο, επιτύχουμε το στόχο που προσπαθούμε να επιτύχουμε αναμειγνύοντας αυτά τα δύο προβλήματα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα το κάνουμε και να ε, γίνονται τα πράγματα ξεκάθαρα, διότι αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε όπως πρέπει. Παρατήρηση δεύτερη. Η προσέγγιση της κυρίας Πλάμ και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, στη γνωμοδότηση όντως όπως είπατε ε, το φύλλο, τη γεωγραφία και τη γενναία. Το πρόβλημα της γυναικείας φτώχειας επιδεινώνεται σε κάποια γενναία η οποία έχει πληχθεί από τη φτώχεια, διότι πρόκειται ακόμα για μια γενιά η οποία δεν κατάφερε να ενταχθεί με ισότιμο τρόπο στην αγορά εργασίας, πρόκειται για μια γενιά η οποία δεν υποφελήθηκε από τα κινήματα ισότητας ε, στην επαγγελματική της ζωή και πρόκειται για μία ε, γενιά η οποία ε, γυράσκει αργότερα. Ε, πρόκειται λοιπόν για ένα πρόβλημα για τις ε, προηγούμενες γενναίες οι οποίες αυτή τη στιγμή πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια και θα δράσουμε πολύ πιο γρήγορα. Το επόμενο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σε επιστήσω την προσοχή κυρία Τσίμερ είναι ότι από γεωγραφική σκοπιά υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες σίγουρα είναι πολύ πιο ε, αποδυναμωμένες ε, σε θέματα φτώχειας από ό,τι άλλες. Να σκεφτώ την Ήπεθρο. Ε, αν δείτε πού επικεντρώνονται τα ευρωπαϊκά κοινωνικά ταμεία, θα πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερη προσοχή ε, στις διαφορές μεταξύ του αστικού κόσμου, για τον οποίο υπάρχουν συγκεκριμένε πολιτικές, υπάρχουν ε, συγκέντρωση πιστώσεων και χρεών και ε, τον κόσμο της υπαίθρου, όπου γίνονται πολύ λιγότερα πράγματα. Και θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη όλα τα προβλήματα κοινωνικής προστασίας, διότι πολύ συχνά η κοινωνική προστασία των γυναικών που έχουν αποκλειστεί από την αγορά εργασίας και φτάνουν αυτή τη στιγμή σε ένα χώρο όπου δεν έχουν εργαστεί και ε, συνδέονται ουσιαστικά με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του συζύγου. Καταλαβαίνετε ότι ορισμένες φορές ε, ε, οι γυναίκες, αυτό είναι γνωστό, ε, ζουν πολύ περισσότερο από τους άντρες. Ε, συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά οι χείρε είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πολλοί κόσμοι δεν θέλουν να το λάβει καν υπόψη. Ακόμα και σήμερα ακούω κάποιους άντρες να λέω «δεν αντέχω άλλο να ακούω για τις χείρε. Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό από αυτό που ε, φαίνεται εξωτερικά. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση. Ε, πέραν των όσων μπορούμε να πούμε υπάρχει πραγματικό πρόβλημα και πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες πολιτικές και μάλιστα αποτελεσματικές πολιτικές για την καλοβόνηση της φτώχειας. Προσβλέπω λοιπόν και εγώ στην αγαστή συνεργασία. Madame Lambert, puis Madame η κυρία Λάμπερτ και μετά η κυρία Γιώτοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρκετά φιλετική αυτή η συζήτηση που διεξάγουμε εδώ. Θα συμφωνήσω με πολλά από αυτά που είπε η κυρία Τσίμερ. Ειδικά για την παραγράφο 4. για τους δείκτες των ανέργων νοικοκυριών για το 2000 20 ε, νομίζω ότι είναι πολύ σωστό και θα πρέπει να το ενισχύσουμε. Θα πρέπει όντω να έχουμε φιλόδοξε εθνικέ στρατηγικέ πριν να ξεκινήσουμε μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρατηγική. Επίση, ε, θα συμφωνήσω και με αυτά που είπαμε για τον σύνδεσμο μεταξύ κοινωνική ασφάλιση και τη διάσταση των ε, δύο φύλων. Επίση, θα ήθελα να πω κάτι για τη μετανάστευση. Το είπε και η κυρία Πλάμ. Ε, είπαμε ότι δεν, δεν έχουμε δεν το, δεν το είδαμε το θέμα των ε, γυναικών τόσο πολύ ε, απλώς μόνο για τις δικές τους ανάγκες αλλά πρέπει να δούμε και τι γίνεται με, την, με τις συζύγους όταν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα στην, ε, σε, τέτοιου, σε τέτοιες ομάδες ε, γυναικών. Γιατί τα άνεργα, νοικοκυριά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ένα σημαντικό, ε, ένα σημαντικό, ένα σημαντικός δείκτης για, τις, για τη γυναικεία φτώχεια. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε αυτό είναι βέβαια το πρόβλημα πάντα με τι γνωμοδοτήσει ότι πάντα υπάρχουν πολλοί περιορισμοί ε, και έτσι απλώ ε, σταχυολογούμε κάποια θέματα χωρί να μπορούμε να τα να διευρύνουμε και να συμπεριλάβουμε πολλά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης ε, και εργασιακών δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικά. Να πω επίση ότι, για το, ότι εδώ είναι και ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε πολλούς, με πολλούς τρόπους είναι, γιατί αν δείτε τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε στέγαση και τα προβλήματα που προκύπτουν, η πρόσβαση στην υγεία πάντα αναφέρεται από τουλάχιστον δύο ε, αναφέρθηκε από τουλάχιστον δύο ε, συναδέλφου, αλλά νομίζω ότι και το θέμα τη στέγαση είναι κάτι που θα πρέπει να μην ξεχνούμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιώτοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την ε, κυρία Τσίμερ για τη δουλειά που έκανε. Συμφωνώ όμω με την ε, συνάδελφο ότι θα πρέπει όντω να τονίσουμε την πτυχή, τη γυναικεία ε, στην έκθεση. Θα δώσω και κάποιε πιο συγκεκριμένε έτσι, απόψεις για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την, ε, τον αποκλεισμό των γυναικών και τη φτώχεια. Ε, η κρίση είναι σημαντική και αυτές που πλήττονται από το πρώτες είναι οι γυναίκες. Η κρίση αυτή έχει γίνει και κοινωνική κρίση γιατί πολλά κράτη-μέλη, δυστυχώς και το δικό μου, αποφάσισαν να λάβουν ε, μέτρα τα οποία μειώνουν τις επενδύσεις στο δημόσιο τομέα. Και κυρίω ε, γυναίκε είναι αυτέ που εργάζονται στο δημόσιο τομέα στη Βουλγαρία τουλάχιστον. Οπότε δεν θα πρέπει να μιλούμε μόνο για γυναίκες που δεν έχουν ε, συγκεκριμένο εισόδημα, αλλά πρέπει να δούμε και γυναίκες που δεν μπορούν να ζήσουν σε ένα σπίτι και συγκατοικούν αναγκαστικά με φίλους ή με συγγενείς. Ε, το χάσμα, το μισθολογικό, παραμένει σε ψηλά επίπεδα στην, ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ε, είναι, μιλάμε για ένα 17%. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη έλλειψη κοινωνικής προστασίας από το κράτος. Δεν υπάρχει υποστήριξη για τα παιδιά, δεν υπάρχουν υποδομές παιδικών σταθμών. Οι γυναίκες που είναι μόνες τους, ας πούμε, οι μονογονικές οικογένειες, οι γυναίκες που είναι μητέρες και είναι ε, μόνες τους, δεν λαμβάνουν καμία, κανένα επίδομα, δεν λαμβάνουν καμία προστασία. Συχνά η φτώχεια των γονιών μεταφέρεται και στα παιδιά. Κάτι άλλο που τονίζει η κυρία Τσίμερ είναι οι γυναίκες από μειονοτικές ε, ομάδες που υποφέρουν από διπλή ε, από διπλή ε, που επιτυχάνουν ε, διακριτική μεταχείρισης και φυσικά αυτό πρέπει να το τονίσουμε όσο δυνατόν περισσότερο. Ε, πρέπει να αναλάβουμε λοιπόν τα απαραίτητα μέτρα για να ενισχύσουμε την απασχολησιμότητα και την κοινωνική προστασία των γυναικών, να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει κατάρτιση ε, να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τα ε, κονδύλια που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι γυναίκες από τις μειονότητες ε, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα διαβίου πρέπει να έχουν τα απαραίτητα προσόντα για την αγορά εργασίας και για τις συμβάσεις εργασίας και αυτό είναι ένα θέμα που το γνωρίζει πολύ καλά η Επιτροπή μας οι γυναίκες συνεχίζουν να είναι τα θύματα αυτών των πρακτικών. Το βρίσκουν πολύ δύσκολο να συμβιβάσουν και την επαγγελματική του ζωή και την οικογένεια και εξακολουθούν να είναι θύματα διακριτικής μεταχείρισης στην αγορά. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Ε, νομοθετικά μέτρα εννοώ. Και βεβαίως θα υποβάλω συγκεκριμένες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Euh, madame Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι όντω είναι μια πολύ καλή αυτή η ευκαιρία για να καταλήξουμε σε ένα στεναρό κείμενο και επιτέλους θα πρέπει να κάνουμε κάτι συγκεκριμένα για τις γυναίκες οι οποίες ζουν σε τέτοιες συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Πρέπει όμω να βλέπουμε και την ε, φτώχεια των παιδιών. Εντάξει, να μην τα αναμειγνύουμε όλα, αλλά μην τα ξεχνάμε και όλα. Γιατί η φτώχεια των παιδιών είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με τη φτώχεια των γυναικών. Εντάξει, δεν είναι αυτό το αντικείμενο του κειμένου. Δεκτό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μιλούμε για την εκπαίδευση στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Ε, αυτό επιτρέπει στις γυναίκες να έχουν επιλογές, ώστε να μπορούν να επιλέξουν ποια θα είναι η καριέρα τους αν δηλαδή εξαιρέσουμε το σχολείο, τότε ε, είναι, προφανώς θα αποκλειστεί κάποιος εάν δεν έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση. Πρέπει λοιπόν να βρούμε ποια είναι τα μέτρα εκείνα που θα αποτελεσματικά θα πολεμήσουν την φτώχεια. Πρέπει να δούμε την εκπαίδευση, πρέπει να δούμε και την επαγγελματική κατάρτιση όμως. Πρέπει να δούμε επίσης τι μπορούμε να κάνουμε για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Εάν ε, κάποιος ε, δουλεύει και δεν έχει καμία ε, βοήθεια όταν μεγαλώνει τα παιδιά του, ε, προφανώς ε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Πρέπει να υπάρξει κάποια πρόνοια για αυτούς τους γονεί. Μιλούμε και για μετανάστριες γυναίκες και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Το έχουμε συζητήσει βεβαίως πάρα πολύ. Αν δείτε τις μειονοτικές ομάδες γενικώ, είναι κάτι που επηρεάζει και τις γυναίκες και τα παιδιά κατά επέκταση. Οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε όσο δυνατόν περισσότερο αυτές τις ε, ομάδε. Η κοινωνική προστασία φυσικά είναι ουσιώδου σημασία. Οι γυναίκε που δεν δουλεύουν πρέπει να ξέρουν ότι μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά του, ότι μπορούν να έχουν οικονομική βοήθεια από κάπου, γιατί αλλιώ ζουν σε συνθήκε απόλυτη φτώχεια. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί πρέπει να μείνουν σπίτι μαζί με τα παιδιά του, οπότε και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μα. Και για να είμαι συγκεκριμένη, τι γίνεται με τις απολύσεις. Πολλές φορές αυτά οι κανόνες που ε, ισχύουν γι' αυτό δεν λαμβάνουν υπόψη τις γυναίκες. Ε, πάντως γενικώ το κείμενο είναι πολύ καλό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό μόνο θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους αν έχουν την ευγενή καλοσύνη να υπογράψουν την ε, ε, γραπτή δήλωση 48 για τις ε, ανήπαντρες μητέρες. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Να συμφωνήσουμε ότι θα, θα βρούμε ποιο θα κάνει τι. Έτσι, πρέπει να τα βρούμε μεταξύ μα. Η κυρία Τσίμερ το είπε πολύ καλά. Εμεί θα ασχοληθούμε με τα θέματα γενικώ τη φτώχεια. Τα θέματα των γυναικών φυσικά είναι σημαντικά. Αναφέρθηκε το ή άλλως πολύ. Αλλά όταν φτάσουμε στις τροπολογίες, νομίζω ότι θα ακούσουμε και άλλα για τις μονογονεϊκές οικογένειες, για τις συντάξεις των γυναικών και διάφορα άλλα. Εντάξει, βεβαίω είναι όλα αυτά σημαντικά, αλλά να μην τα μπλέκουμε όλα, να έχουμε και μια δομή. Να κάνω μια πρόταση. Να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε τη δουλειά μας. πρόσφατα συνάντησα μια, ένα δικηγόρο που ασχολείται με θέματα γυναικών και των δικαιωμάτων των γυναικών και μιλούσε για την ε, ιδέα της ε, πλέον ευημερούσας γυναίκας. Νομίζω ότι πρέπει να συνονιθούμε λίγο με την εισηγήτρια. Ίσως να μπορούσε και αυτό να είναι κομμάτι της συζήτησης. Η εισηγήτρια θέλει το λόγο. Euh, Πρόεδρε, να πω απλώς ότι προσυπογράφω απόλυτα την πρότασή σας. Να έρθει σε ακρόαση η κυρία Αλίνη που έχει εργαστεί με πάρα πολύ γνωστούς ε, δικηγόρους, έχει δει πως έχει κατάσταση των γυναικών στα 27 κράτη-μέλη και νομίζω ότι θα ήταν αξιόλογη η συμβολή της στη συζήτησή μας. Ωραία. Θα δω λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ που ε, καταστήσατε λίγο πιο σαφές ότι ε, υπήρξε η συζήτηση και υπήρξε η απόφαση ε, μεταξύ των δύο επιτροπών να συνεχίσουμε έτσι. Εγώ αυτή τη συμφωνία τηρώ. Οι ε, αρμοδιότητες των δύο ε, επιτροπών είναι συγκεκριμένες έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μία συγκεκριμένη έκθεση για τη, γυνα... για τη γυναική αυτόχεια. Είμαστε έτσι σε ένα σημείο τώρα που πρέπει να συμφωνήσουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά. Η δική μας ε, η αρμοδιότητα, το δικό μας το καθήκον είναι να δούμε τα γενικά σημεία, τις γενικές πτυχές και να συμπεριλάβουμε τη δουλειά που έχει κάνει η Επιτροπή Γυναικών στη δική μας. Δηλαδή ε, η, Επιτροπή των Γυναικών δεν θα ψηφίσει υπέρ των δικών μας επιτρο, ε, προτάσεων, θα τις συμπεριλάβει κατευθείαν στην ε, γνωμοδότησή της. Θέματα φύλων, ε, γεωγραφικά, μειονότητες, εθνοτικές μειονότητες, γυναίκες που μεγαλώνουν μόνο τα παιδιά τους. Είναι πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, είναι πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις, κοινωνικές καταστάσεις που πρέπει να τις, ε, να τις καταστήσουμε πιο συγκεκριμένες. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, γιατί όλοι είμαστε εδώ και λέμε ναι, αλλά ξέρουμε επακριβώς τι θέλουμε και τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να συμπεριληφθεί. Ε, ε, εγώ το συμμερίζομαι αυτό που λέτε, αλλά ε, και εγώ θα ήθελα να το κάνω. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να ακούσουμε και μέσω των επιτροπών και της, των ε, ε, ανθρωπολογιών συγγνώμη, και τις υπόλοιπες απόψεις και να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε το κείμενο. Αλλά σας παρακαλώ, καταλάβετε το. Ε, ας μην θεωρήσουμε ότι εμείς ως Επιτροπή Απασχόλησης με, θα, θα, γίνουμε ανόητοι αν κάνουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε να υπάρξει στενή συνεργασία με την Επιτροπή Γυναικών. Θέλουμε μια πολύ καλή, συγκεκριμένη, ειδική και ταυτόχρονα συνεκτική έκθεση για την, για την Ολομέλεια. Για την Ολομέλεια τι θέλουμε. Στην Ολομέλεια θέλουμε να περάσει αυτή η έκθεση ως έκθεση του Κοινοβουλίου, στην οποία, την οποία εμείς επηρεάσαμε. Ε, καταλάβετε το λοιπόν αυτό που λέω, γιατί πραγματικά μπορούμε, δεν μπορούμε να μπούμε τώρα σε όλες τις ε, λεπτομέρειες για τα δικαιώματα των γυναικών. Η, κυρία Λάμπερτ είπε κάτι. Απλώς εγώ να πω ότι ναι, είναι σημαντικό η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός να, να τα δούμε και ως ε, δικαίωμα ε, ανθρώπινο. Φυσικά είπαμε ότι θέλουμε να μιλούμε για επιθετικές ε, ε, λύσεις όταν μιλούμε για κοινωνικό αποκλεισμό και για φτώχεια αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να ζητούμε μεμονωμένα αιτήματα προς, το, προς τα συστήματα τα κοινωνικά εάν δεν δίνουμε, εάν εμείς δικαιώματα ε, θεμελιώδη στα άτομα αυτά. Και αυτό ισχύει για τις γυναίκες. Ας πούμε, ε, ε δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε ε, καθαρό νερό, σε πρόσβαση σε στέγαση που να μπορούν να την ε, πληρώσουν, σε θέρμανση. όλα αυτά χρειάζονται. Γι' αυτό έχω βάλει την αναφορά εδώ στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό η επιχειρηματολογία για την επικουρικότητα όταν θα επιλέξουμε τους δείκτες Εντάξει, το ξεκινούμε από διαφορετικά σημεία όμω. Πρέπει καταρχήν να δούμε τι σημαίνει όταν μιλούμε για ε, μη κοινού δείκτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για τις ε, προτάσεις σας και για τις απόψεις σας, ελπίζω να μπορέσουμε να μετακινήσουμε λίγο τα πράγματα και να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση και με την Επιτροπή των Γυναικών. Σας ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια. Φυσικά τίποτα δεν απαγορεύει στα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών ε, Υποθέσεων να καταθέσουν ε, τροπολογίες απευθείας ε, σε ό,τι αφορά τα θέματα που αφορούν τις γυναίκες απευθείας στην Επιτροπή Γυναικών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την σοφία μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε ό,τι αφορά την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών, θα κλείσει στις 6 το απόγευμα τον Οκτώβριο, στις 6 Οκτωβρίου θα τις εξετάσουμε τον Αύριο στις 9 ε, Νοεμβρίου συγκεκριμένα θα ψηφίσουμε και 29.30 θα αποφανθεί και η Επιτροπή για τα δικαιώματα των γυναικών. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με το σημείο αυτό της μερισιάς διάταξης. Απλά θα ήθελα να δώσω το λόγο για πολύ λίγο στον κύριο Αλεσάνδρο Σέρκας τις διαπραγματεύσεις συγκεκριμένα για την ενιαία άδεια. Ε, Euh, θα ήθελα να μας πει πώς προχωρούν τα πράγματα με το Συμβούλιο πριν ε, μιλήσουμε τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα, για τρία λεπτά μόνο, να σας πω τρία πράγματα. Να σας υπενθυμίσω καταρχάς τι συνέβη, μετά να σας αναφέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και τρίτον να σας πω τι θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες. Να σας υπενθυμίσω καταρχάς τι έχει συμβεί. Στις 15 του μήνα είχαμε μια συνάντηση τριμερούς διαλόγου άτυπου μεταξύ Επιτροπής ΛΥΜΠΕ της Καθήλων Αρμόδιας Επιτροπής του Συμβουλίου Βελικής Προεδρίας δηλαδή και εμού του φαινομένου. Στις 28, αυτή τη βδομάδα δηλαδή, συναντήθηκα με τους σχεώδες συζητητές και πολύ σαφώς τους εξέθεσα την κατάσταση. Τι βρίσκεται πάνω στο τραπέζι. Επιτροπή ΛΥΜΠΕ μόλις ψήφισε την έκθεσή της, που σημαίνει ότι κοντεύουμε, πλησιάζουμε στο τέλος. Θυμίζω ακόμη ότι η έκθεση αυτή έχει αυτό το τμήμα που αφορά την ενιάδεια, η Επιτροπή Λίμπε είναι αρμόδια. Υπάρχει όμως και ένα άλλο τμήμα στην έκθεση αυτή, το οποίο αφορά τα δικαιώματα, τα εργασιακά και τα κοινωνικά εργαζομένων από τρίτες χώρες οι οποίες έρχονται στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση νομίμως και αυτό αφορά τη δική μας αρμοδιότητα. Η οδηγία αυτή ενδεχομένως να λησμονήσει και τα δικαιώματα ισότιμης μεταχείρισης γιατί μένει μόνο στα διοικητικά ζητήματα της ενιαίας άδεια. Η Επιτροπή λοιπόν ΛΥΜΠΕ είναι μεν η κύρια επιτροπή, η καθήλυνα αρμόδια, εμείς όμως που ασχολούμαστε με τα δικαιώματα, έχουμε απλά προσκληθεί να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση. Όπως είπα, κοντεύουμε να φτάσουμε στο τέλος. Η Επιτροπή Λίμπες δεν θα, Λίμπε δεν θα ε, δυσκολευτεί, νομίζουμε, να συμφωνήσει με το Συμβούλιο και σε πρώτη ανάγνωση με το κείμενο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν προβλήματα τα οποία παραμένουν και θα σας αναφέρω τα δύο σημαντικότερα από αυτά. τα οποία, μεταξύ, τα οποία ε, σε παραθέσεις δεν τα έχουμε με την, με, το, με την Επιτροπή την Ευρωπαϊκή τα προβλήματα αυτά. Αύριο μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και να εγκρίνουμε την νομοθετική πρόταση. Το Συμβούλιο δεν δέχεται την νομοθετική πρόταση τη Επιτροπή. Θέλει να την κάνει πιο σκληρή, αν θέλετε. Ποια είναι τα προβλήματα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα κοινωνική ασφάλιση. Μόλι ψηφίσαμε την έκθεση Λάμπερτ για το θέμα αυτό υποστηρίξαμε την απόφαση του Συμβουλίου βάσει της οποίας εργαζόμενοι από τρίτες χώρες ε, που έρχονται σε μια χώρα παραδείγματος χάρη έχουν όλα τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης. Υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί σε σχέση με την προστασία την οικογενειακή ε, που δεν υπάρχουν πλέον. Αν ας πούμε ένας εργαζόμενος από το Βέλγιο πάει στη Γερμανία, την Ισπανία, στην Ιταλία, όταν φτάνει σε μια νέα χώρα τέλος πάντων έχει τα δικαιώματα τη χώρα στην οποία εργάζεται άνευ ε, περιορισμών. Αυτό λέγεται στον κανονισμό 883 και υπάρχει ισότιμη μεταχείριση για τους επικός χωρών. Η ισότητα ε, μεταχείρισης προβλέπει ότι κάποια πράγματα πρέπει να πάνε προς τα πίσω και να λάβουμε υπόψη κάποια θέματα κοινωνικής ασφάλισης ώστε ε, όταν θα έρθουν οι μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχουν αυτά τα δικαιώματα. Εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε το Συμβούλιο να δεχτεί ότι το θέμα αυτό έχει ήδη ε, ληφθεί υπόψη και υπάρχει ισότητα μεταχείρισης για τους μετανάστες που έρχονται από την, ε, ε, εκτός Ευρώπης, ανεξάρτητα από το που ήρθαν. Δεν θέλουμε να επιστοχωρήσουμε. Είναι κάτι το οποίο έχει λυθεί. Επίσης, Υπάρχει θέμα με τους ε, υπαλλήλου από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε ότι αν αυτοί οι εργαζόμενοι καλύπτονται από την ε, οδηγία για τι αποσπάσει, την οδηγία 46, δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην οδηγία νέα μεταχείριση. Αλλά αν δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία 46, θα θέλαμε να του καλύπτει αυτή η οδηγία. Γιατί αλλιώ ε, θα ισχύει η νομοθεσία τη χώρα καταγωγή του, που σημαίνει ότι επιχειρήσει τρίτων χωρών θα μπορούν να αποσπούν εργαζόμενου ε, στην Ευρώπη με μισθού και κοινωνικά δικαιώματα τη χώρα καταγωγή του. Διότι δεν θα καλύπτονται από την οδηγία για τι αποσπάσει και δεν θα καλύπτονται και από την οδηγία της ενίας άδεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και μπορεί να προκύψει στο πρόβλημα σε, ε, στο μέλλον στο κοινοτικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί μαζί μας, αλλά στο Συμβούλιο υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες είναι ε, πολύ αντίθετες σε αυτό. Και για μα εδώ έρχεται η κόκκινη γραμμή. Εγώ μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, μέχρι την Παρασκευή στις 12, δέχομαι ως εισηγητής ε, προτάσεις για τις ε, προτάσεις που μας κάνει το Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, στις επόμενες εβδομάδες θα συνεχίσουμε αυτό τον άτυπο ε, τριμερή διάλογο για να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε πρώτη ανάγνωση σε συμφωνία. Αν δεν μπορέσει όμως να καταλήξει σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η, νομοδότηση, η οδηγία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να αναλύσουμε αναλυτικά όλα τα στοιχεία της οδηγίας και να έχουμε ένα νομοθετικό μέσο το οποίο ε, δεν θα μας οδηγήσει σε ένα κύμα ρατσισμού, σε ένα κύμα διαφωνίας για τους εργαζόμενους που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δικαιώματα. Ε, αυτά τα έγγραφα ενιαίας άδειας ε, θα ήθελα να τα προσέξετε διότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά θέματα δικαιωμάτων και ελευθεριών. Ε, βιώνουμε πάρα πολύ ευαίσθητε εποχέ, το βλέπουμε και σε άλλα θέματα και θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ καλά πώ ε, συμπεριφερόμαστε στου ανθρώπου που μετακινούνται και που έρχονται στην Ευρώπη. Θα πρέπει να υπάρχει ισότητα δικαιωμάτων με του Ευρωπαίου πολίτε. Και ε, επαναλαμβάνω, μέχρι την Παρασκευή στις 12 δέχομαι τις απόψεις σας γραπτός για τις προτάσεις που κάνω στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Euh, Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Θα στείλουμε μια επιστολή στο σύνολο των μελών της Επιτροπής ε, με βάση αυτά που είπατε και πολύ σωστά λέτε και εσείς ότι τα θέματα αυτά είναι ιδιαίτερως ευαίσθητα και το βλέπουμε και στην επικαιρότητα άλλωστε. Νομίζω ότι με βάση την έκθεση που μας κάνατε, την έκθεση της κατάστασης, θα δώσουμε στα μέλη της Επιτροπής μας τη δυνατότητα μέχρι την Παρασκευή να ανταποκριθούν. Ουσιαστικά ολοκληρώσαμε την ημερησιά διάταξη για το σημείο αυτό. Το μόνο που μου μένει πλέον είναι να καλωσορίσω τον Επίτροπο Λάσλο Αντόρ. Είχαμε ήδη κάποιες συζητήσεις ε, πριν μπούμε στην αίθουσα, βλέπω ότι οι συμβουλευτέ μα πριν μπουν στην αίθουσα είχαν κάποιε συζητήσει μαζί του. Ελπίζω να μην εξάτληξαν το θέμα για να μπορέσουμε και στην Επιτροπή μα να συζητήσουμε. Βέβαια, είμαι σίγουρη ότι έχει να μα πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ο Επιτρόπο για το πρόγραμμα εργασία στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου του. Euh, euh, euh, Καλώ ήρθατε κύριε Επίτροπε, τα, και στην κοινή, τα είπαμε και στην κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Λίμπε χθες για την κατάσταση των Ρωμά συγκεκριμένα και αυτά που διακυβεύονται. Σήμερα θα επικεντρώσουμε την συζήτησή μας και εσείς την παρουσίασή σας φαντάζομαι στον προγραμματισμό των εργασιών, ιδίως όπως είπα σε ό,τι αφορά το δικό σας χαρτοφυλάκι και στη συνέχεια θα υποβληθείτε στο... σε κάτι το οποίο αρχίζετε να συνηθίζετε, νομίζω πολύ καλά, σε ερωτήσει των μελών δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, πράγματι όπως είπατε και εσεί, κυρία Πρόεδρε, χθε είχαμε μια συνάντηση η οποία για μένα ήταν πάρα πολύ επικοδομητική. Με βοήθησε να καταλάβω ποιε είναι οι απόψει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με του Ρωμά. και επειδή τα συζητήσαμε χθε θα περικόψω και κάποια κομμάτια από την εισαγωγή που θα έκανα. Σίγουρα παραμένουν πολλά πράγματα να πούμε ακόμη, διότι όπω είπε και ο πρόεδρο ε, στην ομιλία του πριν από κάποιε εβδομάδε ε, για την κατάσταση τη Ένωση στο Στρασβούργο, όπω καταλαβαίνουμε Πρέπει να ενισχύσουμε την απασχόληση στις θέσεις εργασίας αυτή την περίοδο και πολλά πρέπει να γίνουν στον δικό μου τομέα αρμοδιότητας, ε, τις κοινωνικές υποθέσεις δηλαδή και την απασχόληση. Η σημερινή συνάντηση λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή και νομίζω ότι αντικατοπτρίζει ε, την αποφασιστικότητά μας ε, για να έχουμε πολύ καλές σχέσεις εργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Γνωρίζω ότι θα θέλετε ενδεχομένως να συζητήσουμε και κάποια άλλα ζητήματα της επικαιρότητα και όχι μόνο το πρόγραμμα εργασίας. Χθες είχαμε μια διαδήλωση εδώ η οποία μας θύμισε ποια είναι τα καθήκοντά μας. Και νομίζω ότι έδωσε πολύ λαβή για συζήτηση και σκέψη και φυσικά θα υποκύψω στον πειρασμό και θα κάνω κάποια σχόλια παρά το ότι χθες έκανα μια δήλωση για τη διαδήλωση. Σίγουρα πάντως είναι σημαντικό ο διάλογός μας να, είναι, να γίνεται με ανοιχτό πνεύμα. Γιατί ο κοινωνικός ε, διάλογος είναι σημαντικό στην Ευρώπη και αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του, του κοινωνικού μοντέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι διτές. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα άμεσα βραχυπρόθεσμα προβλήματα, τα οποία χρειάζουν ε, λύσεις για να βγούμε από την κρίση. Και ιδίως σε ό,τι αφορά την βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ένας πιο μακροχρόνιος ορίζοντας. Έχουμε και άλλες μακροπρόθεσμες προκλήσεις, προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ε, την γέρωση του πληθυσμού, την παγκοσμιοποίηση, την αλλαγή του κλίματος. Όλα αυτά σίγουρα απαιτούν ε, μακρόπνες διαρθρωτικές αλλαγές και θα πρέπει όλα αυτά να τα αναλύσουμε αλλά και να ε, δούμε λίγο προβλεπτικά τι μέλη γενέστε και να προσαρμοστούμε στις αλλαγές. Εάν θέλουμε να διαχειριστούμε τις διαδικασίες και όχι μόνο να είμαστε απλοί παρατηρητές και παθητικά αντικείμενα, θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε τα συστήματα κοινωνικής προστασίας των χωρών μας. Εξού και συγκροτήσαμε και χαράξαμε μια νέα στρατηγική για τα επόμενα χρόνια, την Ευρώπη 2020 δηλαδή, για e, ευφυή απασχόληση και δημιουργία θέσεων εργασία. Στην απασχόληση στι κοινωνικέ υποθέσει ε, σίγουρα δίνεται σημαντικός ρόλος. Το 2011 το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν θα αφιερωθεί κυρίως στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020. Εγώ στο δικό μου χαρτοφυλάκιο βλέπω τρεις βασικές προτεραιότητες για το επόμενο έτος. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η αλληλέγγυα ανάπτυξη, να γίνει πραγματικότητα. Δηλαδή να δημιουργήσουμε κατεπηγόντω περισσότερε θέσει εργασία, αλλά να ε, παράσχουμε και υποστήριξη ειδικά για τι ευάλωτε ομάδε. Γι' αυτό λοιπόν και στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 υπάρχουν κάποιε εμβληματικέ πρωτοβουλίε και κάποια σημαντικοί στόχοι. Και η κοινωνική πολιτική με την απασχόληση διαδραματίζουν στι περισσότερε από αυτέ πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Μία έχει να κάνει με την απασχόληση, μια άλλη με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη φτώχεια. Και αυτό πραγματικά αποτελεί ένα ιστορικό επίτευγμα. Με βάση την εμβληματική πρωτοβουλία ε, την ε, νεολαία σε κίνηση που εγκρίθηκε στι 15 Σεπτεμβρίου, η προτεραιότητά μας τώρα είναι να βελτιώσουμε την εκπαίδευση των νέων, επομένω την απασχολησιμότητά τους και την πρόσβασή τους σε ποιοτικέ θέσεις εργασίας. Επιπρόσθετα, πριν τα τέλη του τρέχοντος έτους θα παρουσιάσω και ένα νέο θεματολόγιο για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη ε, σημασία στην έννοια τη ευελιξίας με ασφάλεια και των δεξιοτήτων. Επίσης θα δούμε και την ε, μετάβαση σε μια ε, κοινότητα, πιο, σε μια κοινωνία μάλλον πιο οικολογική, με λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Και θα έχουμε και τις σχετικές προτάσεις για τον κοινωνικό αποκλεισμό. Του χρόνου επίσης ε, με την αλληλέγγυα ένταξη θα συνεχίσω να υποβάλλω προτάσεις αλλά και για την καταπολέμηση της στόχης του κοινωνικού αποκλεισμού. Αγαπητοί βουλευτές, τον επόμενο μήνα η Επιτροπή θα διατυπώσει τις πρώτες της ιδέες για την ε, αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το επόμενο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα παρουσιάσουμε το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους. Είναι σαφές ότι οι ανάγκες ε, που έχουμε για δαπάνες θα πρέπει να κατοπτρίζουν τις ε, προκλήσεις που έχουμε ως Ένωση και θα πρέπει να βοηθούν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Άρα θα πρέπει να βάλουμε τα χρήματα εκεί που θα μπορούν να έχουν τη μεγαλύτερη προσθέμενη αξία. Το βασικό μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του, να στηρίζει την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη στενή διασύνδεση αυτού του ταμείου με την Ευρώπη 2020 στο μέλλον. Θα πρέπει να ξαναδούμε το σύστημα παράδοσης ε, και να είναι προσανατολισμένο πιο πολύ προς τα αποτελέσματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο νομίζω θα πρέπει να προβάλλεται περισσότερο, είναι πιο ορατό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τα χαράς λοιπόν να έρθω και στο αμφιθέατρο του, της Ολομέλειας την επόμενη εβδομάδα, μου το ζητήσατε, και να μιλήσω για το πολύ κρίσιμο αυτό θέμα. Έχω δει ήδη το σχέδιο ψηφίσματος ε, της Επιτροπής σας και μπορώ να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι χαίρομαι που βλέπω ότι η ανάλυση και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγεται για τις βασικές παραδείγματος χάρη αποστολές και δραστηριότητες του ΕΚΤ, τους κανόνες κτλ. Οι απόψεις μας συμπίπτουν αρκετά. Το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση επίσης έχει διαδραματίσει ένα σπουδαίο ρόλο ε, ως ανταπόκριση στην κρίση. Γνωρίζετε ότι και αυτό είναι ένα ταμείο που συνδέεται στενά με το ΕΚΤ. Το 2009 διευρύναμε το πεδίο εφαρμογή για παρεμβάσεις για να μπορέσουμε να στηρίξουμε απολυμμένου εργαζομένους ε, λόγω της κρίσης. Αυξήθηκαν οι αιτήσει και γι' αυτό ε, φαίνεται ότι χρειαζόταν τελικά αυτή η υποστήριξη. Στο πλαίσιο του προγράμματος εργασία μας για του χρόνου θα προτείνω την επέκταση ε, των παρεκκλήσεων που σχετίζονται με την κρίση μέχρι το 2013, αν και λήγουν το 2011. Επίσης, σκοπός είναι να παρουσιάσω ένα νέο EGF για μετά το 2013 ε, για πιο αποτελεσματικούς ε, μηχανισμούς ώστε να φτάνουν ε, οι πόροι γρηγορότερα στους απολυθέντες εργαζομένους. Δεύτερη προτεραιότητα, οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος των δημογραφικών αλλαγών. Η γύρανση του πληθυσμού πραγματικά έχει πολύ μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, ε, ιδίω για το εργατικό δυναμικό, για την υγεία, για την περίθαλψη και για τα συνταξιοδοτικά συστήματα. Η πράσινη βίβλος για τις συντάξεις ε, που παρουσιάσαμε τον Ιούλιο ουσιαστικά δρομολόγησε μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τους κοινωνικούς εταίρους για το μέλλον των συνταξιοδοτικών μας συστημάτων. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημασία έχει το ζήτημα της βιωσιμότητας των συντάξεων, της επάρκειας των συντάξεων να μπει στο πολιτικό θεματολόγιο και να δούμε πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει στην εκπλήρωση ε, των στόχων και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων. Το θέμα είναι περίπλοκο και σχετίζεται με τη διαγενειακή αλληλεγγύη σε στιγμές κρίσης που πραγματικά ε, δημιουργούν προβλήματα και περιορίζουν τον κοινοτικό προπολογισμό. Θέλω να ακούσω και τι απόψει των μελών τη Επιτροπή σα και του Κοινοβουλίου. Όταν λοιπόν ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσει, θα πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Εγώ βλέπω ότι χρειάζεται και μία λευκή βίβλος για να ανταποκριθούμε στις απόψεις που θα διατυπωθούν και για να διατυπώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Τρίτη προτεραιότητα. Δικαιώματα εργαζομένων και πολιτών η κατάσταση, η δεινή των ε, Ρωμά ε, θα παραμείνει ε, στην ημερήσια διάταξη για την Κομισιόν. Βέβαια κάποιες λεπτομέρειες τις είπαμε χθε. μπορώ λοιπόν να παρακάψω αυτό το σημείο και αν υπάρχουν ερωτήσεις μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερο λεπτομεριακά την ένταξη των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κοινωνία. Πριν ολοκληρώσω, αγαπητοί βουλευτέ, θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για το συνεχιζόμενο έργο τη αναθεώρηση τη εφιστάμενη νομοθεσία για τη σωστή εφαρμογή και επιβολή τη. Ένα από του σημαντικού τομεί είναι το εργατικό δίκαιο, η εργασιακή νομοθεσία, που φαντάζομαι ότι σα ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Πρώτα απ' όλα, οδηγία για το ωράριο εργασία τελευταία απόπειρα αναθεώρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως γνωρίζετε, ε, κατέληξε σαν διέξοδο. Από την ε, πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από νομικής ούτε από πολιτικής πλευράς δεν είναι μια κατάσταση που θα τη χαρακτήριζα βιώσιμη. Ο πρόεδρος Μπαρόσο ανέλαβε μια δέσμευση σχετικά και την οποία θα ε, τηρήσω και εγώ. Πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή και να ακολουθήσουμε μια νέα προσέγγιση για το ωράριο εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν αλλαγέ ε, στα εργασιακά πρότυπα. Αυτά θα, οι αλλαγέ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη νέε εξελίξει στι τεχνολογίε των πληροφοριών και των επικοινωνιών πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να προετοιμαστούμε προσεκτικά. Το Νοέμβριο θα ξεκινήσουμε διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Θα είναι η δεύτερη φάση των διαβουλεύσεων και θα υποβάλουμε μια έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας αλλά και μια μελέτη για τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των κανόνων για το ωράριο εργασία. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ξεφύγουμε από το σημερινό αδιέξοδο και εγώ θα κάνω πάντα δυνατόν για να καταθέσω νέες προτάσεις ε, στο πρώτο εξάμεινο του 2011. Νέες προτάσεις που να μπορέσουν να προσφέρουν αποδεκτές προς όλους λύσεις. Ένα άλλο εξίσου δύσκολο νομοθέτημα είναι η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Υπάρχουν δύο είδη προβλημάτων. Πρώτον, προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας. Δεύτερον, πώς θα βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων αφενός και των θεμελιωδών ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς αφετέρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την ουσία του θέματος αυτή τη στιγμή και τον τρόπο με τον οποίο θα υποβάλει τι προτάσει τη. Έχει ξεκινήσει λοιπόν το προπαρασκευαστικό έργο θα πρέπει να έχουμε διαβουλεύσεις με μια ευρία γκάμα ενδιαφερομένων φορέων, μεταξύ αυτών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Κοινωνική Εταίρη και μετά να εγκρίνουμε την πρότασή μας. Και αυτό δεν προβλέπεται να συμβεί πριν το τελευταίο τρίμηνο του 2011. Ξέρω μου βουλευτές, εγώ είμαι υπέρ μιας ισχυρής κοινωνικής διάστασης στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η αρχή η οποία διέπει τις ε, πράξεις μου και τις ενεργές μου. Διότι τελικά δεν προσπαθούμε ε, με την πολιτική να γεμίζουμε ε, τα αρχεία μας ε, με θεωρίες και θεωρητικά πράγματα, διότι υπάρχουν πολίτες οι οποίοι είτε άμεσα είτε έμεσα πλήττονται, υποφέρουν από την χρηματοοικονομική, τη χρηματοπιστωτική κρίση. Υπάρχουν εργαζόμενοι με πάρα πολύ κακέ ε, συνθήκε που φοβούνται ότι θα απολυθούν από τη μια μέρα στην άλλη ή που ήδη έχουν χάσει τη δουλειά του. Υπάρχουν επίση νέοι που δεν μπορούν να βρουν δουλειά, που έχουν πάρα πολύ δύσκολε, ε, ε, πολύ μικρέ δυνατότητε να σταδιοδρομήσουν. Είναι κάποιοι που είναι κοντά στην ηλικία τη συνταξιοδότηση που φοβούνται για τι συντάξει του. Και ξέρω ότι συμμερίζεστε τι ανησυχίε μου και είμαι πεπισμένο ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά για να βελτιώσουμε τα πράγματα από κοινού. Και τώρα θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας ιδέες για όλα αυτά που σας είπα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Έχετε μεγάλη επιτυχία βλέπω γιατί παρά τα πηγαδάκια, τις ιδιωτικές συνομιλίες που είχατε πριν από τη δημόσια ε, συνεδρίασή μας εδώ υπάρχουν 16 συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν το λόγο. Θα εφαρμόσουμε λοιπόν ε, κανόνε ώστε να μπορέσουν όλοι να λάβουν το λόγο. Πριν όμω δώσω το λόγο στου συναδέλφου, θέλω απλά να σα πω ότι σε ό,τι αφορά την πράσινη βίβλο για τι συντάξει, γνωρίζετε ότι στην Επιτροπή μα ε, διερωτηθήκαμε για το κατά πόσον μπορούμε και εμείς ε, να, να το κάνουμε όπως όλοι. Να σεβαστούμε δηλαδή την προθεσμία που έχετε ορίσει για τη δημόσια διαβούλευση. Σε ό,τι αφορά όμως το Κοινοβούλιο, θα έχετε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου μετά από τη Σύνοδο της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2011. Και ελπίζω να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε το δικό μας ε, χρονοδιάγραμμα στο δικό σας για την προετοιμασία των επόμενων ε, σταδίων. Θα δώσω πρώτα απ' όλα το λόγο στους συντονιστές για τρία λεπτά. Ο Γη λοιπόν πρώτα και Θέρκας μετά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόσεξα ιδιαίτερα τα όσα μας είπε ο Επίτροπος και εξ όσων βλέπω ε, σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο για τα θέματα τουλάχιστον απασχόλησης ε, και κοινωνικών θεμάτων, διότι και εμείς στην Επιτροπή μας άλλωστε με αυτά ασχολούμαστε. Δεν θα σχολιάσω την παρέμβασή σας, διότι νομίζω ότι όλα λίγο πολύ ήταν σαφή. Ερωτήσεις όμως. Καταρχάς, πώς προχωρά η διαδικασία των συντάξεων τι προσδοκίες έχουμε για την επόμενη χρονιά. Εγώ θα ήθελα να προωθήσουμε λίγο πιο γρήγορα τη διαδικασία, να ε, επιταχύνουμε λίγο το χρονοδιάγραμμα, ε, διότι χρειάζεται χρόνος για να ετοιμαστούν οι εκθέσεις ε, και προβλέπονται και διασκέψεις, ακροάσεις. Θα θέλαμε να μπορέσουμε λοιπόν να εμπλουτίσουμε αυτή τη διαδικασία. Στη χθεσινή συζήτηση για τους ε, αφήγγανους της Ευρώπης προσπαθήσαμε να βρούμε μια συντονισμένη λύση, να προχωρήσουν τα πάντα προς την ίδια ε, κατεύθυνση και εκεί διαπίστωσα ότι υπάρχουν ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο Επίτροπος και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το ζήτημα η Επιτροπή μας. Θα πρέπει να υπάρξει και μια στρατηγική ελέγχου για τη στρατηγική του 2020. Δεν μπορούμε να ξοδεύουμε χρήματα χωρίς κανέναν έλεγχο. Θα πρέπει να γίνουν και αντίστοιχες αναλύσεις για να δούμε αν υπάρχουν επιτυχίες ε, βάσει των προσπαθειών μας. και ελπίζω να προχωρήσουν οι προτάσεις ε, οδηγιών ε, οι οποίες αναφέρεται, διότι θα πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες όλων. Αν κατάλαβα καλά, Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να περιμένουμε για φέτος και ε, θα ήθελα να δω αυτή την πρόταση που μας αναφέρατε για τη Λευκή Βίβλο. Οι ημερομηνίε ήταν αρκετά σαφείς και σε γενικές γραμμές νομίζω ότι αυτά ήταν τα πιο σημαντικά στα οποία ήθελα να σταθώ. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον ίδιο οικοδομητικό τρόπο στο μέλλον και με τον Επίτροπο αλλά και με το Συνέλο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ ο κύριος Θέρκας και στη συνέχεια η κυρία Χάρκιν. Να πω απλά στον Επίτροπο ότι οι συντονιστέ το έχουν συζητήσει. Μιλώ για το χρονοδιάγραμμα διαβουλεύσεων για την Πράσινη Βουλή για τι συντάξει δεν ζητούμε, όπως αναφέρθηκε στην, πρόταση, στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων, αναβολή ε, της προθεσμίας ε, για τις διαβουλεύσεις όπως ε, πρόβλεψε η Κομισιόν. Ενημερώσαμε απλά την Κομισιόν ότι εμείς ε, έχουμε το δικό μας χρόνο και μπορεί να μην συμπίπτει ακριβώς με το χρόνο της δημόσιας διαβούλευσης και φαντάζομαι ότι καταλαβαίνει πολύ καλά αυτά ο κύριος Επίτροπος. Λοιπόν, Θέρκας και μετά Χάρκιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Θα προσπαθήσω μέσα σε τρία λεπτά να παρουσιάσω τρεις ιδέες. Πρώτον, κύριε Επίτροπε, μου φαίνεται πολύ χρήσιμο αυτό που κάνατε εσείς σήμερα. Αναφερθήκατε δηλαδή και στα θέματα της επικαιρότητα, στα θέματα τα οποία ανησυχούν τους Ευρωπαίους πολίτες και δεν ε, σταθήκατε μόνο στο πρόγραμμα εργασίας το δικό σας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της υπηρεσίας σας αλλά ε, την ε, ε, δύναμη που υπάρχει στους δρόμους που την είδαμε χθε. ο κόσμος είναι ζωντανός και παρόν. υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες στους πολίτες. Ελπίζω όλα αυτά να συνεχιστούν ώστε να προβληθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους Ευρωπαίους πολίτες. Εσείς αναλαμβάνετε κάποια θέματα όπως το θέμα των Αθήγανων ε, πραγματικά υπόψη σας και ελπίζω ε, το σύνολο των Επιτρόπων να αρχίσει ε, για πρώτη φορά να έχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι αντίστοιχο με τις ανησυχίες των πολιτών. Τώρα, για το νομοθετικό πρόγραμμα που μας παρουσιάσατε, που νομίζω ότι είναι πολύ λογικό, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και ένα μικρό σχόλιο για την οδηγία για το χρόνο εργασίας. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι το Κοινοβούλιο ήταν πάντα διατεθειμένο να βρει δρόμους που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα διέξοδα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη σε συγκεκριμένα ε, θέματα. Ε, πάντα όμως είχαμε και μία πολύ στεναρή θέση ως προς ένα κριτήριο το οποίο συζητάμε όλοι. Ναι, ευελιξία κύριε Πρόεδρε, αλλά πάντα με ασφάλεια. Το θέμα δηλαδή του flexicurity. Δεν μπορείτε να δώσετε μία απάντηση που θα αναφέρεται μόνο σε απόλυτη ευελιξία χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα, το κοινοτικό κεκτημένο, τη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Εάν επιτευχθεί αυτή η ισορροπία από πλευρά σα, κύριε Επίτροπε, εμεί ω Κοινοβούλιο θα συνεργαστούμε μαζί σα. Και τελευταίο σχόλιο, αυτό που ενδιαφέρει εμένα περισσότερο. Αναφερθήκατε σήμερα σε θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου σα, αλλά εμεί θεωρούμε ότι το πρόβλημα δεν είναι το δικό σα το χαρτοφυλάκιο, ούτε η δική σα δουλειά, ούτε καν η δουλειά των επιτρόπων. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη λαμβάνει αποφάσει. Ε, και από πλευρά ε, συναδέλφων σας, αλλά κυρίως το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο προχωρά μία σειρά από πολιτικές όπου διαπιστώνουμε ότι καταρχάς έχουμε λιγότερη Ευρώπη και τα πράγματα είναι περισσότερο διακυβερνητικά. Το πρόγραμμα του Φαν Ρόμπαϊ ε, φαίνεται να εκπλήσεται κάθε φορά που ζητάμε να συμμετάσχουμε και το ECOFIN φαίνεται να έχει πολύ πιο σημαντικό ρόλο από το ε, ECOSOC υπάρχει ανισορροπία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα που συζητούσαν όλοι χθε στο δρόμο. Αυτό ζητούσε ο λαό χθε στο δρόμο. Ζητούσε να υπάρχει μια ισορροπία και με τα κοινωνικά θέματα. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το άρθρο 9 των συνθήκων. Δεν μπορείτε εσεί να χρησιμοποιείτε το άρθρο 9 των συνθήκων. Αυτό βρίσκεται και στο πρόγραμμα των συναδέλφων σα και στο πρόγραμμα του Συμβουλίου. να υπάρχει δηλαδή πάντα και η οριζόντια ε, ρήτρα που να ανησυχεί και εσάς και τους υπολείπους. Η κυρία Χάρκιν και μετά η κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Και εγώ χάρηκα με αυτά που άκουσα σήμερα το πρωί. Μιλήσατε για την απάντηση στο χτες και στο σήμερα και, από το, και για το ποιες είναι οι επιδιώξεις που έχετε, αλλά θα πρέπει να προσθέσω κάτι. Ε, όλα ε, αυτά ε, βασίζονται στην αρχή ότι υποσχόμαστε να κάνουμε αυτό που μπορούμε και τελικά κάνουμε όντως και αυτό που υποσχόμαστε. Γιατί η πραγματικότητα των, της καθημερινής ζωής των ανθρώπων είναι διαφορετική. Βλέπουμε ποια είναι η, βλέπουν την κατάσταση και περιμένουν από τους πολιτικούς να βελτιώσουν τις, ε, να βελτιώσουν τις συνθήκε ζωή του. Ε, δεν μπορούμε εμείς λοιπόν να μην τηρούμε αυτά που λέμε. Χαίρομαι που βάζετε, που ε, βάζετε στην ίδια ζυγαριά το, την πολιτική για το 2020 με το ESF, με το Κοινωνικό Ταμείο. Ξέρω ότι προσπαθούμε, προσπαθούσαμε να ε, πείσουμε τους Ιρλανδούς να ψηφίσουν ναι στην συνθήκη τη Λισαβόνα και πολλέ αφήσει έλεγαν ε, υπόσχονταν δουλειέ, δουλειέ, δουλειέ και σήμερα μα ρωτάνε πού είναι τελικά όλε αυτέ οι δουλειέ. Πρέπει οι πολίτε να ξέρουν πώ μπορούν να συμμετάσχουν, πώς μπορούν, ποια είναι, ποιες είναι οι ευκαιρίε που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν ε, τη ζωή του. Ε, πρόκειται να ε, δημιουργηθεί το νέο ταμείο από το 2013 και μετά. Ας δούμε όμως τι γίνεται μέχρι τότε και ας βασιστούμε βεβαίω και στα διδάγματα που θα έχουμε για, το μετά το 2013. Μιλήσατε για τη μακροπρόθεσμη πρόνοια όταν είπατε για δημογραφικές αλλαγές. δεν είπατε όμως τίποτε για... Δεν είπατε λίγο περισσότερε πληροφορίες γι' αυτό. Τι ακριβώ εννοείται με τη μακροπρόθεσμη πρόνοια. Επίση, υπάρχει η νομοθεσία και πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί καλύτερα. Γιατί αυτό, είπαμε, έχει επίδραση στις ζωές των ανθρώπων. Και συμφωνώ με τον κύριο Σέρκας ότι μιλούμε για την ε, ισοτιμία μεταξύ των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων των εργατών και των θεμελιωδών ελευθεριών της αγοράς. Μιλήσατε για το άρθρο 9. Ναι, αλλά οι εργαζόμενοι δεν βλέπουν, ε, δεν, δεν συνδέουν τις, δεν συνδέονται με τις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες της αγοράς, συνδέονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι δικά τους. Ε, νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Συμφωνώ με αυτό που λέτε, ότι όταν υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων, υπερασπιζόμαστε και τα δικά μας δικαιώματα. Αυτό που μας είπατε σήμερα είναι πολύ ε, φιλόδοξο και φυσικά ε, προσβλέπω στην ε, συνεργασία μας. Λάμπερτ και μετά Τσίμερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για την παρουσίασή του. Πρέπει να παραδεχθώ κύριε Επίτροπε ότι θαυμάζω την αισιοδοξία σας ότι μπορούμε να βρούμε λύση για το ωράριο εργασίας. Συγκριτικά όμως σε ό,τι αφορά ε, τη μετάβαση σε μια οικονομία ε, με, χαμηλή, με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, μάλλον θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Ε, και έχουμε και το θέμα ε, των θέσεων εργασίας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ απαραίτητα, όπως είπατε. Και εκεί, ε, μάλλον στο θέμα του ωραρίου εργασίας, αναφέρατε και τις ε, διάφορες νέες μορφές απασχόλησης που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι ε, υπάρχουν ε, στην ε, πρόταση για το ωράριο εργασία υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία δεν είναι πολύ ξεκάθαρα, νέε τεχνολογίε, φροντιστέ. Πρέπει να δούμε πώ μπορούμε όλα αυτά να τα εντάξουμε κάπου. Ένα συνάδελφο που δεν μπόρεσε να παραστεί μου ανέθεσε να σα κάνω μια ερώτηση σε σχέση με την γονική άδεια, την άδεια πατρότητα συγκεκριμένα. Γνωρίζουμε εσείς και η κυρία Ρέντινγκ πιστεύετε ότι δεν μπορεί να μπει στο, στα θέματα της άδειας μητρότητας. Ε, θα ήθελα να ε, επαναλάβετε ότι έχετε τη δέσμευση, ε, ότι θα κάνετε μια ξεχωριστή πρόταση, θα λάβετε μια ξεχωριστή ε, απόφαση, μια ξεχωριστή πρωτοβουλία το 2011 για την άδεια πατρότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και τώρα συζητούμε την ε, οδηγία για την άδεια μητρότητα. Κάτι άλλο το οποίο μα ενδιαφέρει είναι πώς βλέπετε να εντάσσεται η συνέχιση της κοινωνικής πολιτικής ε, στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Έχουμε την πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά βέβαια ε, η κοινωνική ε, πολιτική δεν αφορά μόνο τα θέματα της καταπολέμησης της αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ άλλων και πραγματικά θα μας ενδιέφερε να δούμε τις προσπάθειές σας. Ξέρω ότι σωστά αποδίδεται προσοχή αυτή τη στιγμή ε, στην πολιτική καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω καταγωγής, φιλετικής κτλ. Αλλά θα θέλαμε γενικώ να προωθήσετε τις προτάσεις αυτές και την ε, εφαρμογή τους. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική και την ε, μερίσια διάταξη για την ένταξη, την, ε, την ενεργό ένταξη, active inclusion, πώς θα συνεργαστείτε με επιτρόπους από άλλες γενικές διευθύνσεις για να προχωρήσουμε και με τις δημόσιες υπηρεσίες ε, που θέλουμε να είναι ποιοτικές και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, και για την ε, μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. κυρία Τσίμερ και μετά θα απαντήσει στις πέντε πρώτες ερωτήσεις ο Επίτροπος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπε η Τζιν Λάμπερτ για το αισιοδοξία και για την ε, πρότασή σα που θα, ότι θα υποβάλλετε νέα πρόταση για το ωράριο εργασία. Ε, κι εγώ πλάγιν. Ε, μήπως ο πρόεδρο Μπαρόσο δεν ήταν που είπε, που ότι άλλαξαν οι καιροί και θα πρέπει να, το νέο ωράριο να, αντικατο, να αντικατοπτρίζει αυτές τις αλλαγές. Ε, αυτό όμως γιατί γίνεται για την αλλαγή της ε, παραγωγικότητας, για τη μείωση των ανώτατων ορίων των ορών εργασίας. Θα περιμένουμε βεβαίω να δούμε ποια θα είναι η πρότασή σας, αλλά νομίζω ότι θα πάει στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θέλετε. Επίσης, άλλα μερικά σχόλια ακόμη. Ε, θέμα της ε, χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ως Επίτροπος ε, Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόληση, θεωρώ ότι έχετε την ευθύνη να ασχοληθείτε και με το θέμα αυτό. Γιατί μιλούμε για κοινωνικά δικαιώματα που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων και κάποια από τα μεμονωμένα άρθρα δεν έχουν επικυρωθεί ακόμη μέχρι σήμερα. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να μας πείτε εσείς, σε συνεργασία και με άλλους συναδέλφους σας, πώ θα δραστηριοποιηθείτε στον τομέα αυτό, ώστε να μπορέσετε να συμβάλλετε, ώστε να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο τη χάρτα. Επίσης, Μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της φτώχειας του κοινωνικού αποκλεισμού, την οποία θα παρουσιάσετε φέτος το, το, μέχρι το τέλος του έτους. Ε, θα, μου, θα μου άρεσε να μου πείτε ακριβώς πώς θα το παρακολουθήσετε αυτό, δηλαδή κάτι άλλο πέρα από μια εκστρατεία για την αποδοχή στην, ε, της, ε, στην κοινωνία, τι ακριβώς θα κάνετε ώστε να έχουμε δηλαδή συγκεκριμένα εργαλεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει συγκεκριμένα εργαλεία ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει τα θεμελιώδη δικαιώματα στα κράτη-μέλη. Μιλώ κυρίως για το πρόβλημα που υπάρχει σε συνεργασία και με, τους, ε, με τον Επίτροπο για θέματα ενέργειας. Όταν δηλαδή μιλούμε για μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ή για την, ε, ε, για την καλύτερη ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Και από την άλλη πρέπει να βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη αποφασίζουν το κόστος αυτής της ε, νέας, αυτών των νέων υποδομών να μετακυλίονται στους ενοικιαστές ή στους κατόχους των σπιτιών. Ε, δεν πρέπει να κάνουμε να υπάρχει μια κεντρική πολιτική. Δεν είναι στην ατζέντα μας δηλαδή η χρήση, η ηλεκτρική ενέργεια, η πυρηνική ενέργεια. Τι κάνουμε με όλα αυτά δεν πρέπει κι εσείς μεταξύ σας ως ε, επίτροποι να ε, συντονιστείτε. Η πρόεδρος διακόπτει την κυρία Τσίμερ. Κυρία Τσίμερ, συγγνώμη, αλλά ξεπέραστε κατά πολύ το χρόνο. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο να απαντήσει. Μένουν άλλες 10 ερωτήσεις. Ελπίζω να μην σπαταλήσετε τα 40 λεπτά που απομένουν για να απαντήσετε στις πρώτες 5 απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να απαντήσω στι περισσότερες από τι ερωτήσει ε, που ετέθηκαν σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα των διαβουλεύσεων για τι συντάξει. Δεν θα ήθελα να παρατείνουμε την επίσημη περίοδο που λήγει στις 15 ε, Νοεμβρίου, αλλά ε, έχω την πεποίθηση ότι θα ακουστεί φωνή του Κοινοβουλίου. Εάν γίνει βέβαια αυτό όπως είπατε, ε, είπατε για Φεβρουάριο του 2011 εσείς. Εάν δεν πάμε τόσο μακριά στο επόμενο χρόνο, φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη τις απόψεις του Κοινοβουλίου όταν θα ξεκινήσουμε τις προετοιμασίες μας για το follow-up, που όπως είπα μάλλον θα είναι μια λευκή βίβλος, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσουμε στο δεύτερο τρίμηνο. Θα ήθελα να κινηθούμε λοιπόν και να εργαστούμε βάσει αυτή τη διερευνητική ε, προθεσμία, αυτό το διερευνητικό χρονοδιάγραμμα που σας παρουσίασα για να λάβουμε υπόψη και τις δικές σας ε, συνεισφορές. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να εμείνουμε στην επίσημη προθεσμία γιατί όλοι οι υπόλοιποι εμπειρογνώμονες, ε, οι ομάδες πίεσης θα μας στείλουν ε, τις ε, απόψεις τους μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε όλες αυτές τις πληροφορίες. Θα ήθελα επίσης να πω ότι έχουμε τον Οκτώβριο στις 29 του μήνα συγκεκριμένα ε, μια συνεδρίαση, μια συζήτηση για την Πράσινη Βίβλο. Θα είστε κι εσείς βέβαια ευπρόσδεκτοι και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε έναν πάρα πολύ επικοδομητικό διάλογο με την Επίτροπο. Δεν το ανέφερα, ε, θα το πω τώρα. Υπάρχουν κάποια θέματα σε ό,τι αφορά την υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία. Θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση στο MRI. Χθε συναντήθηκα με κάποια μέλη ε, του Κοινοβουλίου και κάποιους άλλους εμπλεκόμενους φορείς στο Κοινοβούλιο εδώ και σας επιβεβαιώνω ότι πριν τα τέλη του έτους θα διατυπώσουμε νομοθετική πρόταση μετά την ολοκλήρωση της ε, μελέτης επιπτώσεων. Νομίζω ότι μπορούμε να τηρήσουμε αυτή την ε, προθεσμία. Και η διαδικασία νομίζω ότι μετά θα είναι αρκετά δυναμική Θα έχουμε μετά και μία πρόταση για τις μυοσκελετικές διαταραχές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε και την πρόταση για την έκθεση ε, στον καπνό του τσιγάρου. Και φυσικά και θα ακούσουμε τις δικές σας ε, απόψεις, γιατί το Κοινοβούλιο έχει έναν απαραίτητο ρόλο να διδραματίσει τον τομέα αυτό. Κάποια ακόμη ζητήματα που θα ήθελα να σχολιάσω για τα, γιατί ετέθησαν από συναδέλφου σα. Ξεκινώ με το ρόλο της ε, ευελιξίας με ασφάλεια και της πολιτικής απασχόλησης. Πώς θέλουμε εμείς να διαμορφώσουμε τη συζήτηση στο μέλλον, με ρωτήσατε. Δεν μπορώ να προδικάσω το πλαίσιο του θεματολογίου αυτού σίγουρα μια νέα προσέγγιση για την έννοια flexicurity θα υπάρχει και μια νέα προσέγγιση για την έννοια της κινητικότητας, κάτι που ξεκίνησε με την πρωτοβουλία νεολαία σε κίνηση. Αυτή την που είναι σε την εμβληματική, όπως τη λέμε, πρωτοβουλία. Θέλουμε να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη, για παράδειγμα, τον επιμικημένο επαγγελματικό βίο τις διαφορές που υπάρχουν στις ανάγκες και στις δεξιότητες των διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Η ευελιξία δεν αφορά μόνο τους νέους. Ε, όσο περισσότερο άλλες ηλικιακέ ομάδες οι οποίοι ε, θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που δίνει αυτό το πρόγραμμα Flex Security για μετάβαση από μια θέση απασχόληση σε μια άλλη. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας ε, στις ανάγκες των καιρών, διότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ και θα επηρεάσουν βέβαια την ουσία της πρότασης και άλλες σχετικές ε, πρωτοβουλίες. Η επιτυχία των πρωτοβουλειών μας μεταξύ αυτών και οι στόχοι 2020 θα βασιστούν, θα εξαρτηθούν από την διακυβέρνηση. Με τη Βελγική Προεδρία γίνεται σημαντική δουλειά. Ο ρόλος του Συμβουλίου ΕΦΣΚΟ, ο πιθανός μηχανισμός παρακολούθησης της πρόοδου στο μέλλον, πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε ακόμη, και το λέω με ειλικρίνεια, διευθετήσει τα, πάντα τα πάντα. Προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε τον απαραίτητο ρόλο και την ε, απαιτούμενη βαρύτητα σε αυτούς οι οποίοι επηρεάζουν τις πολιτικές απασχόλησεις και κοινωνικών θεμάτων. Προσπαθώ να είμαι συνεπής ό,τι αφορά τις ε, δεσμεύσεις μας και την υλοποίησή τους. Φυσικά και υπάρχουν πράγματα για τα οποία θέλω να είμαι αισιόδοξο και μεταξύ αυτών είναι και το θέμα του ωραρίου εργασία. Συμμετείχα στον πρώτο γύρο ε, των διαβουλεύσεων του κοινωνικού εταίρου. Πράγματι, είναι γεγονό ότι δεν είναι όλε οι συναντήσει που έχουμε μαζί του ενθαρρυντικέ. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι για παράδειγμα οι συναντήσεις που έχω με εκπροσώπους ε, της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν ότι υπάρχει μια νέα προσέγγιση, ένα μεγαλύτερο άνοιγμα από πλευράς τους. Άρα θα πρέπει να αναζητήσουμε, να επιδιώξουμε κάποιες νέες προσεγγίσεις, νέες λύσεις. Υπάρχει χώρος, νομίζω, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε έστω και λίγο αισιόδοξοι. Σίγουρα πρέπει να αφήσουμε χώρο στους κοινωνικούς εταίρους να διατυπώσουν τις δικές τους προτάσεις, να εκφράσουν ε, τις ενδεχόμενες νέες ανάγκες τους εάν ε, έχουν σχέση με τις προτάσεις μας και βέβαια περιμένω να ανακύψει και μια νέα δυναμική μετά τη δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών για την αξιολόγηση δηλαδή του κοινωνικού οικονομικού πλαισίου και για την εφαρμογή της οδηγίας. Νομίζω ότι όλα αυτά θα δώσουν μια νέα διάσταση στο διάλογο. Ίσως μάλιστα οδηγήσουν και κάποια, σε κάποιες εξελίξεις, σε κάποια νέα βήματα. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για τις αποσπάσεις εργαζομένων, τη συζήτηση για τα κοινωνικά δικαιώματα, όταν επεξεργαστούμε αυτά τα θέματα και καταλήξουμε σε μια πρόταση θα περιλαμβάνεται σίγουρα η αναφορά στο κοινωνικό δικαίωμα και δι στο δικαίωμα της απεργίας. Δεν φαντάζομαι ότι θα μπορούσαμε να καταθέσουμε μια πρόταση που δεν θα περιλάμβανε αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών πτυχών. Και στόχος μας βέβαια είναι να έχουμε μια καλύτερη οδηγία που θα έχει καλύτερα αποτελέσματα, όχι μια οδηγία που θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερες ε, αντιπαραθέσεις και αυτό σίγουρα θα ήταν επιζήμιο. Το παράδειγμα των ε, σχεδίων ενεργειακής απόδοσης, το οποίο αναφέρθηκε, είναι ένα ζήτημα που πραγματικά μπορούμε να επεξεργαστούμε με άλλους επιτρόπους, όπως ε, τον κύριο Έτιγκερ για παράδειγμα. Υπήρξαν συζητήσεις, ε, πραγματικά δεν έχουμε διερευνήσει απαρκώς το τι μπορούμε ακόμη να κάνουμε. Διότι η κατάσταση διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Υπάρχουν κράτη που κάνουν πολλά σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά αυτά έργα έχουν σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο καθότι μειώνεται το κόστος της ενέργειας για τα νοικοκυριά. Μπορούμε λοιπόν να επεξεργαστούμε τέτοιες προτάσεις και στη συνέχεια να προβούμε και ε, σε επανακαθορισμό της ε, του σχετικού θεματολογίου και θα συνεργαστώ με τον ε, αρμόδιο επίτροπο. Σε ό,τι αφορά την άδεια πατρότητας, το έχω ξαναπεί. Είναι θέμα της Αντιπροέδρου Ρέντινγκ, ξεκάθαρα και φυσικά και θα τις αναφέρω το ενδιαφέρον το οποίο εκφράσατε. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ακούσουμε δύο ακόμη πεντάδες ομιλητών. Δυστυχώς θα σας παρακαλέσω να περιοριστείτε ο καθένας στο ένα, άντε στο ενάμιση λεπτό. Ο κύριος Μπακ και μετά ο κύριος Ντερός. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε ε, Επίτροπε, να σας ευχαριστήσω για τα λόγια σας, για τα καλά σας λέω για το συνδικαλιστικό κίνημα και τα όσα είπατε για το κοινωνικό, την κοινωνική πτυχή της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, επειδή πιέζει ο χρόνος, ένα σημείο θα ήθελα να θίξω το οποίο έχει να κάνει και με μία από τις προτεραιότητές σας, την ε, ε, ανάπτυξη, συμμετοχική ανάπτυξη. Ε, θέλετε να εξασφαλίσετε θέσεις εργασίας, είπατε, και θα ήθελα να μιλήσω για τα προβλήματα που υπάρχουν στο δίκτυο Eures. Από το 1993 υπάρχει το δίκτυο Eures για την προώθηση και ενίσχυση των, ε, της διασυνοριακής κινητικότητας. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο λοιπόν ε, στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Euros όμως δεν ε, αφορά μόνο την, ε, ε τις θέσεις εργασίας αλλά και την ε, κοινωνική ασφάλιση, θέματα φορολογικά. Η Κομισιόν τώρα, ε, χωρίς κάποιο λόγο, μείωσε την ενίσχυση του Euros και έχει ε, περιορίσει και τον αριθμό των ε, συμβούλων. Ε, για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό κύριε Επίτροπε, συμφωνείτε μαζί μου ότι αυτό, το, αυτή η κατάσταση είναι ιδιαίτερος άσχημη ε, κυρίως για κάποιες συνοριακές περιοχές. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσετε την ενίσχυση του εργαλείου αυτού με τα ίδια κονδύλια για την οδηγία για τις ε, αποσπάσεις και την οδηγία για την ε, εργασία. Χαίρομαι για τις ε, διαπραγματεύσεις που κάνατε με τους, νέους, με τους κοινωνικούς εταίρους και φαντάζομαι ότι με, τις, βάση τις έρευνες που έγιναν θα έχετε και νέα στοιχεία. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Uh, thank you, Ευχαριστώ τον Επίτροπο που είναι σήμερα εδώ. Δύο πράγματα γρήγορα. Και στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο γίνεται λόγος για το ότι πρέπει να λαμβάνεται η υπόψη ε, η αίσθηση της ε, αγοράς. Ναι, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και την αίσθηση που έχουν οι άνθρωποι που ε, διαδήλωναν χτε στις Βρυξέλλες και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή εμπειρία είναι λίγο πικρή. Αυτό μας είπαν κάποιοι συνδικαλιστές από την Ιρλανδία χτες που έχουν παλέψει χρόνια για την ε, στρατηγική της Λισαβόνας. Να μην ε, αγνοούμε λοιπόν τους κινδύνους, οπότε σας ρωτώ, εσείς τι συμβολή έχετε, η γενική σας διεύθυνση τι συμβολή έχει να δώσει στις προτάσεις που υπάρχουν για την οικονομική διακυβέρνηση. Δεν βλέπω κανένα σημείο στις έξι προτάσεις που ακούστηκαν χτες ότι υπάρχει οποιοδήποτε οικονομική σκέψη ή κοινωνική σκέψη σε αυτές τις ε, ε, προτάσεις. Δεύτερον, οι κοινωνικές υπηρεσίες. Εγώ είμαι εισηγητής, αν ε, ξέρετε για το θέμα αυτό. δεν είναι σαφές απόλυτα, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό των εγγυήσεων όσων περιγράφονται από πολλούς ως ο πυρήνας της κοινωνικής Ευρώπης. Εγώ είμαι υπέρ μιας ε, πολυτομιακής task force, μιας ομάδας κρούσης με εμπειρογνώμονε, με ενδιαφερόμενου, υπό την ηγεσία τη Κομισιόν βεβαίω, κατά πάσα πιθανότητα και από τη δική σα διεύθυνση, που θα καταγράψει ποιε είναι οι αλλαγέ που πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό. Γιατί Υπάρχουν, υπάρχουν πολλές έρευνες εκθέσεις που, που λένε πρέπει να γίνει αυτό και το άλλο θεωρητικά, αλλά δεν υπάρχει δράση. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Η κυρία Λίν και μετά η κυρία Μωράν. Ε, yes, thank you very much. Κυρία ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που αναφερθήκατε στην εφαρμογή και επειδή αναφέρεστε και στην εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων αλλά και τις υπόλοιπες οδηγίες, θα ήθελα να ξέρω αν έχετε κάποια πράγματα επιπλέον να μας πείτε γι' αυτό. Όσον αφορά τώρα τις δημογραφικές αλλαγές, ε, και πάλι με χαροποιεί το γεγονός ότι μία από τις βασικές σας πρωτοβουλίες αφορά τις δημογραφικές αλλαγές. Και θα ήθελα να ξέρω αν έχετε κάνει κάποιε περαιτέρω συζητήσει για τον κώδικα διοντολογία. Ε, Όπω ξέρετε, έχω παρουσιάσει και σχετική προφορική ερώτηση και το ψήφισμα που ε, ψήφισε το Κοινοβούλιο επί του θέματο. Επίση, ε, την πράσινη βίβλο για τι αποζημιώσει. Το συζητήσατε και στο παρελθόν. Ετοιμάζεται κάτι καινούργιο από αυτού. Επίσης, ε, ε, την ηλικία συνταξιοδότησης. Το πότε κάποιος λαμβάνει τη συνταξιοδότησή του, ε, αλλά το κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε μία υποχρεωτική ηλικία στην οποία κάποιος θα σταματάει να εργάζεται. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εργαστούν αργότερα, ε, περισσότερα χρόνια και να ε, θέλουν να λάβουν τη σύνταξή τους αργότερα. Θα το λάβουμε αυτό υπόψη. Επίσης, ε, είδα ότι ασχολήθηκε με τα θέματα του χρόνου εργασίας και την οδηγία. Ελπίζω να είστε και εσείς αισιόδοξους και να πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση από το τους. Και χαίρομαι που ε, κάναμε και όλες αυτές τις συζητήσεις για τους Ρωμά εχθές και σας ευχαριστώ που ήσασταν στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ μαζί μας αυτή την ε, σύνοδο εργασίας. Τρία ερωτήματα θα ήθελα να σας υποβάλω. Καταρχάς, μιλήσατε για ένα νέο ταμείο ευρωπαϊκό ανάπτυξη, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Πώς πιστεύετε ότι θα προχωρήσετε στον εξορθολογισμό για μεγαλύτερη προβολή και καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων όπως έχουν τα πράγματα σήμερα με τα κονδύλια. Υπάρχουν πολλοί πόροι, πολλά μέσα και μηχανισμούς έχουμε στη διάθεσή μας. Ξέρουμε όμως ότι οι εταίροι μας επί τόπου όταν πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν όλα αυτά κάπως ε, τα χάνουν, για να μην πω τα χάνουν πολύ. Πώς μπορούμε λοιπόν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Δεύτερο ερώτημα, πώς μπορούμε να προβάλλουμε καλύτερα τη δράση των ταμείων αυτών επιτόπου και αυτό έχει να κάνει και με το ερώτημα της ε, συναδέλφου Χάρκιν. Πράγματι, ε, είναι σημαντικές οι πολιτικές μας, πολύ λίγο όμως ορατές. Πώς μπορούμε να τις προβάλλουμε περισσότερο στον πολίτη ώστε να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη. Τρίτο ερώτημα τι νέα στρατηγική μπορείτε να προτείνετε σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μετά το 2013. Πώς θα συνδέσετε και την ομάδα εργασίας τη σχετική. Γιατί θα θέλαμε όλοι να συμβάλλουμε στον εξεχρονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου αυτού. Είπατε ότι θα δώσετε τη μάχη της απασχόλησης. Αυτό το ταμείο είναι ένα από αυτά τα εργαλεία. Euh, ο κ. Τούρινεν και μετά θα απαντήσει ο Επιτροπός. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνεχίσω από κάτι που είπε ο κύριος Ντερόσα που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και το είχα σημειώσει και εγώ για να σας ρωτήσω εάν η πρώτη σας προτεραιότητα είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και να διασφαλίσετε ε, ότι θα έχουμε ανάπτυξη ε, και όντως θα καταφέρετε σε αυτή την ε, ε, προτεραιότητά σας, θα έχουμε καλύτερη ανάπτυξη για τις οικονομικές πολιτικές και τις κοινωνικές πολιτικές. Με εξέπληξε το γεγονός εχθές ότι δεν είχαμε καμία αναφορά στην απασχόληση, απλώς έχουμε πολύ μικρή κατανόηση των οικονομικών εξελίξεων και των κυρώσεων. Πώ εσεί, ε, ως Επίτροπος Αρμόδιο για θέματα τέτοια θέλετε να διασφαλίσετε ότι η απασχόληση θα είναι το κλειδί και θα είναι στο επίκεντρο του ε, το που κάνουμε σε οικονομικό επίπεδο. Εγώ ασχολούμαι με θέματα ανέργων, κυρίως ε, νέων ανέργων και ε, θέματα ποιότητας εργασίας και κοινωνικού ντάμπινγκ. Υπάρχουν κάποια προβλήματα και το είδαμε και στην οδηγία για τις αποστάσεις, αλλά υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα και ελπίζω να υπάρξει μια πρωτοβουλία για τις αποσπάσεις. Ελπίζω να ακούσω κάποια πράγματα και από εσά σήμερα γι' αυτό. Χρειαζόμαστε ένα ευρύτερο πλαίσιο για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη, ε, καταπολέμηση της ένδυας ε, και καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ, διότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ελπίζω εσείς ε, και η Επιτροπή μας να θεωρήσουμε το 2011 ως τη χρονιά αφετηρίας συνεργασίας μας σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά τώρα τη στρατηγική το 2020, ε, παρακολουθώ αυτό το θέμα στενά και ελπίζω πολλές ε, από τις ε, προτάσεις μας να συμπεριληφθούν. Σας ευχαριστώ που έχετε περιλάβει κάποια στοιχεία. Δεν βλέπω κάποια πράγματα όμως στο πρόγραμμα εργασίας επ' αυτού. Ο Επίτροπος. Οικονομική διακυβέρνηση. Πράγματι, είναι σημαντικό θέμα αυτό, όχι μόνο για το δικό μου το χαρτοφυλάκιο, αλλά για το χαρτοφυλάκιο της όλης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης διακυβευόταν, το μέλλον του ευρώ διακυβευόταν και έπρεπε να γίνει κάτι για να μπορέσουμε να επαναθεμολιώσουμε τις βάσεις της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, αλλά για μένα αυτό σήμαινε και ενίσχυση των βάσεων της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θεωρώ ως κάτι εξελίξη. Έχουν γίνει κάποια βήματα Έχουμε τρεις ανακοινώσεις ήδη, αλλά όπως ε, σας είπα είναι κάτι το οποίο είναι εξελίξει. Έγινε κάποια πρόοδος για να ε, κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τις ανισορροπίες που υποσκάπτουν τη σταθερότητα του ευρώ και υποσκάπτουν και τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο από οικονομική σκοπιάς αλλά και από πολιτική σκοπιάς. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι ότι τώρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το φάσμα των ανισορροπιών. Δεν αφορούν μόνο την οικονομία αλλά και τα χρέη. Και στο έγγραφο το οποίο παρουσιάστηκε υπάρχει μια πρόταση να εξετάσουμε τα θέματα αυτά όχι μόνο εκ των υστέρων αλλά και εκ των προτέρων. Πρόληψη δηλαδή. Αυτό είναι πρόοδο. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά φυσικά δεν είναι το παν. Ε, μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι κάθε φορά που συζητάμε ε, συμμετέχουμε σε συζητήσεις μακροοικονομικής διακυβέρνησης, κάθε φορά που συμμετέχω εγώ τουλάχιστον, κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου προκειμένου να εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι να συμπεριληφθεί και η ανεργία. Να θεωρείται ένα πολύ σημαντικό θέμα ε, όταν συζητάμε τις μεγάλες ανισορροπίες της οικονομίας. Γι' αυτό και πριν από δύο εβδομάδες ήμουν στο Όσλο για να συμμετάσχω σε μια κοινή συνεδρίαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας διότι αυτή η πρωτοβουλία που ξεκίνησε στην ε, ε, πρώτη τέτοια συνεδρίαση που είχαμε μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, δεν είχαν ξανασυναντηθεί ε, τα δύο αυτά όργανα από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Συγγνώμη, μάλλον δεν πρέπει να μιλάω για τον πόλεμο. Αλλά ήταν ιστορική η συνάντηση αυτή. Ο Ντομινίκ Ροσκάν προείδρευε και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ο κ. Σομάρια, και αυτό που με εξέπληξε ήταν ότι οι συνάδελφοι στο ΕΚΟΦΕΝ δεν ήταν καλά ενημερωμένοι επί του θέματος. Ε, έκανα λοιπόν ότι περνάει από χέρι μου για να το γνωστοποιήσω το γεγονός αυτό, διότι καταρχάς έχουμε την αγορά εργασίας, ε, τα θέματα της πλήρους απασχόλησης, ε, της κοινωνικής ένταξης, της αξιοπρεπούς εργασίας και από την άλλη έχουμε τη μακροοικονομική σταθερότητα. θα πρέπει λοιπόν αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα να μιλήσουν μεταξύ τους και να κατανοήσουν αλλήλους. Όπως σας έλεγα, είναι έργο εν αλλά δεν είναι επικίνδυνη αυτή η αποστολή, ούτε αδύνατη διότι υπάρχει μια σοβαρή δέσμευση για τους στόχους του 2020. Όλοι θέλουν να εμπλακούν σοβαρά και να φτάσουμε πράγματι σε αυτό το 25% ε, που προσπαθούμε να επιτύχουμε και δεν ε, μας ενδιαφέρουν μόνο οι πολιτικές για την αγορά εργασίας αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα διαρθρωθούν οι μακροοικονομικές πολιτικές. Γι' αυτό και βασίζομαι στη δική σας υποστήριξη και στην ε, ε, συμμετοχή σας ε, στις μελλοντικέ συζητήσεις. Τώρα, για τα ταμεία. Όταν μίλησα για ένα νέο ταμείο για την παγκοσμιοποίηση, μιλάμε για ένα ανανεωμένο ταμείο για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση και θέλουμε φυσικά να χρησιμοποιήσουμε την παλιά μας εμπειρία. Ορισμένες φορές ε, ακόμα και ο τύπος μας βοηθάει, διότι μας επισημαίνει κάποιες ελλείψεις δεν διαβάζω μόνο εφημερίδες. Έκανα μια ε, συνάντηση προσφάτως στο Στρασβούργο με τον κύριο Πόρτας, ο οποίος είναι ο ε, εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση και διάβασα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έκθεσή του. Και συμφωνώ μαζί του στο εξή. Ακόμα και αν τελειώσει η κρίση πριν, μετά από ένα-δύο χρόνια, καλό θα ήταν να μείνει αυτό το κατόφλι των 500 για να καθορίζουμε τα πόσον κάποιος είναι επιλέξιμο στο μέλλον. Ακόμα και αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας με δυναμικό τρόπο, θα πρέπει να προβλέπουμε και απώλειες θέσεων εργασίας, εάν ε, υπάρχουν ε, μεταφορές επιχειρήσεων, αν υπάρχουν ε, αντίθετα αποτελέσματα σε εμπορικές συμφωνίες, για παράδειγμα, και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την ε, προσαρμογή στην ε, παγκοσμιοποίηση και να υπάρχει αυτό το κατόφλι, γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε και διευκολύσεις για κάποια κράτη-μέλη. Θα μειωθεί η δυνατότητα του, της κάθε χώρας να αντιμετωπίσουν τις απώλειες θέσεις εργασίας και θα πρέπει να υπάρχει ένα αποτελεσματικό μέσο που να λειτουργήσει ως λίγο ταχύτερα από ό,τι στο παρελθόν και ε, να καταδείξουμε σαφώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η προστιθέμενη αξία σε αυτό το τομέα. Έχουμε κάποιο χρόνο να το επεξεργαστούμε το θέμα αυτό και σας ευχαριστώ για τα όσα μας δώσατε και θα μας δώσατε επί του θέματος. Τώρα, για την εφαρμογή και τις κατευθυντήριες γραμμές. Πριν από κάποιες εβδομάδες ο κύριος Χιούς μου έγραψε για μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που ήθελαν να ασχοληθούν με θέματα ατυχημάτων ε, και κοιτάμε να δούμε αν υπάρχει καλή εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών. Είμαι ανοιχτό σε προτάσεις και θα δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Για τον κώδικα διοντολογίας, ε, όπως σας είπα, εγώ είμαι ανοιχτό στο θέμα αυτό, αλλά τώρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις δημογραφικές ε, τάσεις. Θα το συζητήσουμε την επόμενη χρονιά και νομίζω ότι πρόκειται για μια νέα δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία εγώ θέλω να ενισχύσω και άκουσα με χαρά ότι οι επόμενες δύο προεδρίες και η Ουγγαρία και η Πολωνία ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για να ε, προωθηθεί το θέμα της δημογραφικής αλλαγής και να θεωρηθεί η προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο βασικός λόγος, δεν θα σταθώ σε όλα τα αίτια αυτή τη στιγμή, ο βασικός λόγος για τον οποίο πρέπει να ασχοληθούμε με τα δημογραφικά ζητήματα είναι σε συνέχεια των όσων κάνουμε για τις συντάξεις καθώς επίσης ε, και για την ε, ε, ενεργό γύρανση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και ε, πολιτικές για την οικογένεια, ε, μακροπρόθεσμη ιατρική φροντίδα και πώς η μακροπρόθεσμη ιατρική φροντίδα μπορεί να συνδεθεί και με τη συσσόρευση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και την καλύτερη διαβίωση αυτών που ασχολούνται με τον τομέα. Επίσης, είναι και μια καλή ευκαιρία για θέσει εργασία, αλλά νομίζω ότι αυτό το έχουμε συζητήσει. Το δημογραφικό ζήτημα λοιπόν είναι αναδυόμενο τομέα. και ελπίζουμε ότι σύντομα θα είναι στρατηγικός τομέας. Ε, εάν ληφθεί η σχετική απόφαση θα δούμε και τι γίνεται με την αλικία συνταξιοδότησης. Ε, εάν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν πιέσεις να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης και κάνουμε διάκριση μεταξύ της ε, που κάποιος σταματά να εργάζεται και της ε, ίδιας της ηλικίας συνταξιοδότησης. Θέλουμε να μην υπάρχει πολύ εκτεταμένη χρήση της πρόορης συνταξιοδότησης. Ε, δεν ξέρω αν κάποιος έχει πρόθεση να αλλάξει την ε, ηλικία συνταξιοδότησης. Ε, δεν ξέρω τι γίνεται με το θέμα στη Γαλλία, το ξέρω ότι συζητάτε. Αλλά σίγουρα δεν θα γίνει κάποια ενιαία πρόταση. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά που υπάρχει στα συνταξιοδοτικά συστήματα, στα μοντέλα της αγοράς εργασίας και δεν νομίζω ότι κάποιος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει τοπικές ιδέες και θέλει να κάνει πρόταση για ενιαία μοντέλα. Θα πρέπει να δούμε λίγο ε, και το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικές συνταξιοδοτικές δομές. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ Γκρούνι, και μετά το Μασμάν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Δύο ερωτήσεις ε, έχω. Πάντοτε σχεδόν διαβάζουμε για τη φτώχεια ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πώς θα προωθήσετε τη χρήση του Ταμείου για την καταπολέμηση της φτώχειας. Δεύτερον, γίνεται πολλής λόγος για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και την εξέβρεση ε, θέσεων απασχόληση. Η διατήρηση όμως είναι εξίσου σημαντική. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν να μας πείτε αν θα υπήρχε ενδεχόμενο να λάβετε μια νομική πρωτοβουλία και για την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία σε σχέση με το γεράσκοντα πληθυσμό, ε, απασχόληση ατόμων με αναπηρία, απασχόληση ηλικιωμένων. θα θέλαμε να δούμε τι γίνεται στις επιχειρήσεις, στο περιβάλλον των επιχειρήσεων και ε, θα ήθελα να πείτε αν ε, αυτό το έγγραφο, είπατε για τις μεσοκελετικές διαταραχές ότι θα έχουμε ένα έγγραφο, αλλά ένα άλλο θέμα που επανέρχεται και είναι σημαντικό είναι το στρες στην εργασία. Καθώς και η πρόληψη των αυτοκτονιών στο εργασιακό περιβάλλον που δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε λύση ακόμη πλησματική. Θα ήθελα να μου πείτε επ' αυτόν. Τόμας Μαν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, είπατε ότι έχετε συναντήσει τους ε, κοινωνικούς εταίρους. Μπράβο, πολύ καλά κάνατε, είναι πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε συμμάχους, αλλά έχετε πάρει χρόνο να δείτε και όσους ε, επηρεάζονται από αυτές τις αρνητικές ε, συνέπειες της κρίσης. Εγώ χτες στη διαδήλωση συνάντησα κάποιους από τους ε, από εκπροσώπους ε, ε, εταιριών κατασκευών στη Γερμανία που μειώνονται οι θέσεις εργασίας τους, που απολύονται. Μήπως θα, πρέπει να συνεργαστείτε με τον Επίτροπο Ανταγωνιστικότητας. Μέχρι πού ανοίγουν οι πόρτες σας και πόσο εδίκοα είναι τα ότα σας στα προβλήματα των ανθρώπων αυτών. Επίσης, είναι σημαντικό να, σκεφτώ, να σκεφτόμαστε να, να συνδυαστικά Έχουμε την ε, πράσινη βίβλο για τις συντάξεις. Και έχει καταστεί σαφές πόσο σημαντικό είναι η Κομισιόν να έχει μία φωνή ε, και να μιλά και σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι νέοι άνθρωποι με προοπτική τη σύνταξη. Δεν θέλουμε να έχουμε αγώνα, μάχη μεταξύ των γενεών. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι και κλείνω που μια ε, αίτηση η οποία υπάρχει, ένα αίτημα που υπάρχει μέσα στην ε, έκθεσή μου και η οποία υπερψηφίστηκε σήμερα ε, συμπεριλαμβάνεται και στην δική σας πρόταση. Χαίρομαι λοιπόν που μιλάτε και εσείς στην πρότασή σας για τον ενεργό γύρανση μέχρι το 2012. Ευχαριστώ. Η κυρία Κίνγκα Κούνς και μετά ο κύριος Μπάκα. Köszönöm szépen. Én is Θα ήθελα και εγώ να σας διαβεβαιώσω, κύριε Επίτροπε, για την υποστήριξή μας, διότι θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται οι κοινωνικές πτυχές στις αποφάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει αρκετή ενσωμάτωση των πτυχών αυτών αν δημιουργηθούν θέσει απασχόληση δεν μπορούμε όμως να πετύχουμε την οικονομική ανάκαμψη. Επίσης δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποφύγουμε τον κοινωνικό διάλογο. Πρέπει να πω επίσης ότι σήμερα ε, υπάρχουν παγίδες. Ε, αν χαθεί η κοινωνική διάσταση ε, θα αποτύχουμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι άλλο, κύριε Επίτροπε. Τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα, είναι διατεθειμένα να συμπεριλάβουν τις πτυχές αυτές και στις πολιτικές τους. Δηλαδή θα έχουν κοινωνικό διάλογο, θα έχουν διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Χθε είχαμε τη διαβούλευση για τους Ρωμά. Φυσικά και καλό είναι να γνωρίζουμε δείκτες, χρειάζεται παρακολούθηση οι πόροι που διατίθενται πρέπει να φτάνουν στις περιφέρειες ε, και δει τις ε, μειονεκτικές, ε, τις περιοχές που ζουν άτομα που είναι σε μειονεκτική θέση που ζουν σε απομακρυσμένους διάσπαρτους οικισμούς για παράδειγμα. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά πολλές φορές όταν ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα, ένα έργο, χάνονται, χάνεται η συνέχεια που είχαν αυτά τα έργα. Η κυρία Μπλοκ. Ο κύριος Κλάρκ. Ε, θα επανέλθω στο ερώτημα που σας είχα θέσει την πρώτη φορά που ήρθατε εδώ για τη βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ε, απασχολούν το μισό εργατικό δυναμικό στην Ένωση. Ε, τότε δεν μπορούσατε να μου δώσετε συγκεκριμένα στοιχεία. Τώρα μπορείτε. Ήδη έχετε δώσει συγκεκριμένα στοιχεία σε άλλες περιπτώσεις. Σήμερα το πρωί η Επιτροπή μας ε, ενέκρινε ε, δαπάνες για την ε, υποστήριξη εταιριών που κλείνουν και μετεγκαθίστανται. Ε, ωραίο όλο αυτό, αλλά η ε, εργαζόμενοι. Προφανώς είναι και αυτοί, είναι, δεν, δεν είναι μόνο οι εταιρείε που έχουν ανάγκη για υποστήριξη, είναι και οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι που έχουν ανάγκη να, να τους στηρίξουμε για να μπορούν και αυτοί να στηρίξουν τις οικογένειε τους. τελευταία, στην τελευταία ε, σύνοδο στο Στρασβούργο είπε και ο κύριο ε, Μπαρόσο ότι οι μικρομεσαίες ε, εταιρείε στραγγαλίζονται. και ταυτόχρονα εγκρίνουμε μια έκθεση η οποία έχει μια ρήτρα η οποία προτείνει ε, υπέρογγες εκθέσεις και άχθος διοικητικό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, τι γίνεται. Πριν από λίγους μήνες ψηφίσαμε να αποκλείσουμε τους ε, ανεξάρτητους ε, ιδιοκτήτες φορτηγών από την σχετική οδηγία. Με κάποιο τρόπο αυτό το ξαναείδαμε και τον Απρίλη άλλαξε η ψήφος και η Ολομέλεια ακολούθησε βεβαίως. Τι θα κάνετε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κύριε Επίτροπε. Δεν θέλω φιλοδοξίες, θέλω συγκεκριμένες και λογικές δεσμεύσεις. Η κυρία Πλάμπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο και να τον ευχαριστήσω και για τις απαντήσεις που προσπαθεί να δώσει σε πολύ σημαντικά ε, προβλήματα. και κυρίως τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις συντάξεις. Εχθές με μέλη της πολιτικής μου ομάδας ε, ήμασταν στη διαδήλωση στις Βρυξέλλες, μιλήσαμε με πάρα πολλούς ανθρώπους, άντρες και γυναίκες και μεταξύ των ανθρώπων με τους οποίους συζητήσαμε μου έθεσαν ερωτήσεις ε, για το θέμα αυτό το οποίο δημιούργησε την κρίση και που έχει πολύ σημαντικές κοινωνικές συνέπειες και η ερώτηση ήταν τι μέλη γενέστε και θα ήθελα και εγώ να διαβιβάσω την ερώτηση σε εσά πώς θα αντιμετωπίσετε τις μισθολογικές ε, αποκλίσεις και τις διακρίσεις σε θέματα φύλους, ε, στα θέματα της εργασίας, ε, διότι κατ' εμέ αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα και θα πρέπει να ε, μεταλαμπαδευτούν και στις εθνικές νομοθεσίες. θα πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένη στρατηγική κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του επί του θέματος. Ε, τι σκοπεύετε να κάνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ κύριε Επίτροπε να σας θέσω κάποια ερωτήματα. Μιλήσατε χθε για την οικονομική διακυβέρνηση, διακυβεύονται πολλά. Αλλά κάποιοι ξεχνούν ότι ο όρος οικονομική διακυβέρνηση περιλαμβάνει και την απασχόληση. Κύριε Επίτροπε, στι ε, χθεσινές αποφάσεις ε, του Σώματος των Επιτρόπων δεν είδα τις έξι προτάσει που έχουν τεθεί επιτάπητο. Έξι, έξι φορές αναφέρθηκε το άρθρο 148 τη συνθήκη η νομική βάση. Τώρα, σε αυτή την πολύ σημαντική ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση των Ρωμά. Ε, ακούσαμε τα σχόλιά σας, ακούσαμε τα σχόλια της κυρίας Ρέντινγκ, έχουμε το χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πώς θα αλλάξει αυτό ε, την κατάσταση και τα δεδομένα. Αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα η νέα κατάσταση με, το, με τη συνθήκη της Λισαβόνας ήταν το άρθρο 9. Η χθεσινή απόφαση του Σώματος των Επιτρόπων για την οικονομική διακυβέρνηση ξεκίνησε να θέτει τα εγκάρσια αυτά ζητήματα τα οποία είναι γεγραμμένα στο άρθρο 9 σε ό,τι αφορά την ανάλυση ε, του χρέους το την επιστολή που έστειλε ο κύριος Ρέν στον κύριο Χέντερς. Ποια είναι η διασύνδεση μεταξύ οικονομικών, υπουργών οικονομικών και οικονομίας και υπουργών κοινωνικών υποθέσεων. Και τέλος. Μπορείτε να φανταστείτε ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο όπου το μόνο εργαλείο που θα έχει στη διάθεσή του για να παρέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αποτελεσματικότητα στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση θα εξαφανιζόταν. Merci. Uh, let me start with uh, Λοιπόν, να ξεκινήσω με μία από τις ε, πρώτες ερωτήσεις. Δεν το απάντησα. Είναι μεγάλη ανησυχία και για μένα αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή να ε, το απαντήσουμε διότι τώρα φτάνουμε στις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό και ε, νομίζω ότι θα μπορούσατε να με στηρίξετε κι εσείς ίσως να υποστηρίξετε τον προϋπολογισμό που θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού. είναι πολύ σημαντικό οι πρωτοβουλίες ε, που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να περιλαμβάνει και την ε, πρωτοβουλία για τις ε, θέσεις απασχόλησης για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό το δίκτυο Eures πολύ καλύτερα από ό,τι πριν. Τώρα, για τα ταμεία για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την καταπολέμηση της ένδυας και της ε, δυνατότητες καταπολέμησης της ένδυας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πρόκειται όντως για πολύ σημαντικό θέμα και η Βελγική Προεδρία τον επόμενο μήνα, τον Νοέμβριο δηλαδή, θα οργανώσει μία διάσκεψη η οποία θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη ε, στο θέμα αυτό και θα συμμετέχω κι εγώ και φυσικά θα ακούσω πάρα πολύ προσεκτικά τις απόψεις που θα εκφραστούν στο συγκεκριμένο φόρουμ. Σκοπεύουμε να προβάλλουμε καλύτερα το θέμα αυτό, ε, καλύτερα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θέλουμε να δώσουμε πιο σαφείς προσανατολισμούς από πλευράς πολιτικής. Τι προγράμματα μπορούμε να ετοιμάσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ, σημαντικά, ε, πολύ συχνά συγγνώμη, στις συζητήσεις για τους Ρωμά αναφέρονται πράγματα. Ε, εγώ εχθές ας πούμε αναφέρθηκα στην έννοια στην παρουσίασή μου, διότι ε, δεν είναι μόνο τα ποσά αυτά που έχουν σημασία, αλλά το θέμα είναι τι σχεδιασμούς κάνουμε και όπως είπε και η κυρία Γκέντς, εάν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων είναι βιώσιμα και θα μείνουν ε, ακόμα και μετά το πέρας της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε περισσότερη προσοχή, κάποιες καινοτομίες πρέπει να... Ε, επαναφεύρουμε τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου διότι τα πράγματα είναι πολύ περίπλοκα και σε κάποιες περιπτώσεις ε, ε, έχουμε περιπτώσεις χωρίς προηγούμενο. Είναι πολύ δύσκολο να ε, χρηματοδοτήσουμε πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε και νομίζω ότι αυτό απαντά και στην ερώτηση για τους Ρωμά. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Προσαρμογή στην ε, Παγκοσμιοποίηση μπορεί να χρηματοδοτήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εάν η κατάσταση ή η παγκοσμιοποίηση εν γέννη σε ένα συγκεκριμένο χώρο ε, αφορά άνω των 500 ανθρώπων. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να γίνει συνδυασμός ε, μεταξύ των επιπτώσεων λόγω απώλειας θέσεων εργασίας και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα μπορέσουμε να καλύψουμε στις μελλοντικέ συζητήσει και το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να διαδραματίσει κάποιο ρόλο για να διαμορφώσουμε το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση και να δώσουμε δυνατότητε και στι μικρομεσαίε επιχειρήσει να υποφαληθούν το Ταμείο. Ε, συμμετείχα σε μία διάσκεψη για την οργάνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, αλλά τα βασικά θέματα τα οποία συζητήθηκαν εκεί ήταν η συμμετοχή του στον κοινωνικό διάλογο. Και νομίζω ότι αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Είμαι υπέρμαχος του θέματος και ε, έρχομαι εδώ από μια διάσκεψη για τον τομεακό και κοινωνικό διάλογο, στον οποίο και πάλι ε, μπόρεσα να επισημάνω πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κοινωνικό διάλογο. Ενισχύεται και ο ίδιος ο διάλογος. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το διάλογο αυτό για τη διαχείριση της οικονομίας και της διατήρησης του κοινωνικού μοντόλου. Πράγματι υπάρχει έλλειψη ισορροπιών, ε, γεωγραφικές ανισορροπίες ε, Συν της ε, ακούμε από τους διαφόρους ενδιαφερομένους, κυρίως από τα συνδικάτα, ότι στα νέα κράτη-μέλη ο κοινωνικός διάλογος είναι ανεπαρκής και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τον ενισχύσουμε, διότι μπορεί να υπάρχουν ε, συνέπειες, κοινωνική αστάθεια και φυσικά αυτό σχετίζεται και με το κοινωνικό ντάμπινγκ. Κάποιο κοινωνικό ντάμπινγκ νομίζω στον προηγούμενο γύρο ερωτήσεων. Δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε πολλά πράγματα για το κοινωνικό ντάμπινγκ. όσον αφορά ε, τις θέσεις εργασίας, αλλά όσον αφορά την υποστήριξη του διαλόγου, εκεί μπορούμε να κάνουμε πράγματα και θα συνεχίσουμε φυσικά. Βιωσιμότητα θέσεων εργασίας και εδώ εστιάζουμε την προσοχή μας και εδώ ασχολούμαστε και με θέματα αναδιάρθρωσης. Θα γίνει και μια σχετική πρόταση στο εγγύς μέλλον. Πρόκειται για ένα σημείο ε, όπου έχουμε αλληλοεπικάλυψη με τα θέματα βιομηχανίας και θεωρούμε ότι στην ε, μελλοντική πρωτοβουλία για τη βιομηχανική πολιτική το θέμα της ανατεάθρωσης θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Πρόκειται για μια σημαντική αλληλοεπικάλυψη των δύο θεμάτων. Ενδιαφερόμαστε και εμείς γιατί ακριβώς υπάρχει ενδιαφέρον για την βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας και ε, μάλιστα με ένα πιο κοινωνικά ευαίσθητο τρόπο διατήρησης των θέσεων. Η βιωσιμότητα δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα υγείας και ασφάλειας. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να παραμείνουν όλε οι θέσει εργασία και αυτό ισχύει και για κάποιου κλάδου που αρχίζουν να χάνονται. Για παράδειγμα, ε, τα ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβλέψουμε ότι σταδιακά θα αρχίσει να χάνεται στο μέλλον ε, γιατί ακριβώς ε, η πολιτική ανταγωνισμού και οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και των όσων προβλέπονται εκεί θα αλλάξουν. Στόχος είναι να το διαχειριστούμε αυτό κατά τρόπον ώστε ε, να δείξουμε τη δέουσα ευαισθησία και να διασφαλίσουμε ότι οι περισσότεροι από τους εργαζομένους ε, θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να βρουν νέες θέσεις εργασίας ή δυνατόν στον ίδιο χώρο στον οποίο έχασαν ε, την θέση εργασίας που είχαν. αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται συνεχώς. Ε, θα γνωρίζετε ότι ήταν και στο, ε, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Σώματος των Επιτρόπων. Το είχε θέσει ένα κράτος μέλος. Τέλος, οικονομική διακυβέρνηση. Η επιστολή του Επιτρόπου Ρεν ε, προς τον κύριο Ρέιντερς αναφέρθηκε. Μπόρεσα να μιλήσω με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό Μερκέ, ο οποίος ε, ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για αυτή την επιστολή. Λόγω της ευαισθησίας του θέματος και επειδή το γεγονός ότι η έξοδος μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, βραχυπρόθεσμα για να εφαρμόσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Να έχουμε δηλαδή πε, περισσότερες δράσεις τώρα ή θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε την ανάκαμψη. Η κυρία Μιλκέ νομίζω ότι συμφωνεί και αυτή μαζί μου. Θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη για ανάκαμψη και αυτό φυσικά σημαίνει ότι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη στη νέα δομή διακυβέρνηση η οποία θα προκύψει. Θα το συζητήσουμε και με τον πρόεδρο Φανορόμπαϊ, να δούμε τα θέματα της οικονομικής διακυβέρνησης και ε, ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά, ε, διότι είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας. Βασιζόμαστε σε εσά όταν θα έχετε αυτές τις ανταλλαγές απόψεων να φροντίσετε το 148 να συμπεριληφθεί στη βασική νομική βάση για την οικονομική διακυβέρνηση. Η πρώτη ευχαριστώ τους διερμηνείς που ε, πέρασαν λίγο το χρόνο εργασία. Θα τα ξαναπούμε κύριε Επίτροπε ε, ε, την επόμενη εβδομάδα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τις εργασίες μας στις 25 και 26 Οκτωβρίου είναι προσεχή συνεδρίες επιτροπής μας.